Dámy a páni, dámy a páni, Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ας ε, αρχίσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Σας καλωσορίζω όλους. Το πρώτο σημείο στη μερίσια διάταξη έχει να κάνει με τις δικές μου τις ανακοινώσεις σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών. Έχουμε λοιπόν την έγκριση της ημερήσιας διάταξης ε, για τις συνεδρίες του Μαρτίου. Την εγκρίναμε στο πλαίσιο της ομάδας των συντονιστών. Και επίσης ε, εγκρίναμε το να συμπεριλάβουμε την αναφορά 24-27 όσον αφορά την ισπανική τηλεόραση. Το Μάρτιο θα συμπεριλάβουμε πέντε αναφορές, το ΆΕΛΚΕ θα έχει δύο, οι σοσιαλιστές μία αναφορά και ένα κατεπήγον αίτημα, η φιλελεύθερη μία αναφορά και το FTD μία αναφορά και αυτό. Οι γραμματείες των πολιτικών ομάδων θα πρέπει να διευκρινίσουν εν συνεχεία ποιε τελικά θα είναι αναφορέ οι οποίε θα συμπεριληφθούν. Και αυτό θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλο τη σημερινή συνεδρίαση. Εγκρίναμε επίση την αναφορά 33 του 2019 ω κατεπίγουσα αναφορά από του σοσιαλδημοκράτε η κατάσταση στο Stonehenge και θα συμπεριλάβουμε και αυτή την αναφορά στη συνεδρίαση του Μαρτίου. Επίση, οι συντονιστέ συμφώνησαν να συζητήσουν με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια στη συνεδρίαση του Μαρτίου και θα σας δοθούν περαιτέρω πληροφορίες για το ζήτημα αυτό. Συζητήσαμε τη συνεχεία και τη συνεδρίαση που θα λάβει η χώρα στις 2 και έπειτα στις 11 Απριλίου. Εγκρίθηκαν εδώ πέρα κάποιες προκαταρκτικές ημερήσεις διατάξεις και προβλέπεται εδώ πέρα ότι 12 αναφορές μπορούν να συμπεριληφθούν για τις δύο αυτές συνεδριάσεις του Απριλίου. Δύο από το ΕΛΚΑ, δύο από τους Δημοκράτες, μία αναφορά από τους Φελελεύθερους, δύο αναφορές από τους Πρασίνους, δύο αναφορές από την ΚΟΕ και μία αναφορά για το EFDD και δύο αναφορές για το ECR. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να διευκρινίσουν πάλι ποιε τελικά αναφορές θα συμπεριλάβουν στις ημερήσιες διατάξεις του Απριλίου. Εναπόκειται στις πολιτικές ομάδες να αποφασίσουν προτεραιότητές τους και η σχετική προθεσμία είναι το απόγευμα της Παρασκευής αυτής της εβδομάδας. Επίσης, Επίσης, οι αναφορές 80 74 του 2018 5902 του 2018 θα παραμείνουν ανοιχτές. Η αναφορά 930 του 2018 κρίθηκε παραδεκτή. Και η επιστολή για την αναφορά αυτή θα αποσταλεί στην Ισπανική κυβέρνηση καθώς επίσης και στους συναδέλφους από την Επιτροπή Πολιτισμού και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Τώρα, όσον αφορά τα σημεία υπό το Β, δεν καταφέραμε να τα καλύψουμε αυτά. Θα τα καλύψουμε στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών το Μάρτιο. Αυτά όσον αφορά τις πληροφορίες για την σημερινή συνεδρίαση των συντονιστών. και σας προτείνω τώρα να περάσουμε στην επόμενη μας αναφορά 1030 του 2017. Αναφέρονται ο κύριος Ισμαήλ Αντώνιο Λόπες Πέρες, Ισπανικής Ιθαγένειας, και πρόκειται για μια αναφορά που έχει να κάνει με τα προβλήματα στην περιοχή της Γαλλικίας, της Ισπανίας, όσον αφορά την κατάχρηση των πόρων του ΕΤΠΑ σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Καλησπέρα στη Γαλλικία καίγονται τα βουνά. Πάντα καίγονται, χειμώνα καλοκαίρι. Ε, καίγεται το δίκτυο Natura 2000 και επιπλέον οι πληροφορίε που δίνουν ε, οι τοπικέ αρχέ, η κυβέρνηση τη Γαλλικίας είναι πάρα πολύ λίγε. Ε, δεν υπάρχει διαφάνεια ούτε πληροφορίε ε, σε ό,τι αφορά τι καμένε επιφάνειες, τα καμένα εδάφη και ούτε τα λεφτά που ξοδεύουμε για την πυρόσβεση. Ε, δεν, δεν έχουμε πληροφορίες για την αναδάσωση. Γνωρίζετε ε, ποιος ασχολείται με την ε, αναδάσωση των καμένων επιφανειών στην ε, Γαλλικία. Ο ευκάλυπτος, ο οποίος ε, φύεται όπου να είναι ε, και με αυθόρμητο τρόπο. Ε, υπάρχει ένα παλιό δασικό σχέδιο, το οποίο έχει καταπέσει, δεν έχει επικαιροποιηθεί και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να δίνει λεφτά ε, στην κυβέρνηση της Γαλλικίας που δεν κάνει τίποτα για να λύσει τα διαφορετικά προβλήματα των βουνών και που όλα τα τα δίνει μόνο για την πυρόσβεση. Παρά την ε, σημασία των ε, εκτάσεων αυτών στη Γαλλικία, που είναι περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού εδάφους της, της Γαλλικίας, οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν από το 1992 δεν έχουν σαν σκοπό να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των βουνών, ε, των αυτόχθονων δασών ε, που έχουν υποβαθμιστεί ιστορικά και ε, με ρυθμό επιταχυνόμενο. Αυτό το δασικό σχέδιο υπάρχει από το 1992 και θα έτρεχε μέχρι το 2032 40 χρόνια και μιλούσε για μια μέγιστη επέκταση των ευκαλύπτων σε μια έκταση 245.000 εκταρίων. Η πρώτη απογραφή που έγινε ε, το 72-73 ε, έλεγε ότι οι ευκάλυπτοι κάλυπταν 131.181 ε, εκτάρια. Πιο πρόσφατα, στη Γαλλικία, το 2009, ο ευκάλυπτος βρέθηκε ότι είχε καλύψει 433.000 εκτάρια και καθαρών δασών ευκαλύπτων και μεικτών. Το 2016 η επιφάνεια που κάλυπτε ο ευκάλυπτος είχε ξεπεράσει τα 500.000 εκτάρια και μάλιστα 13 ε, χρόνια πριν φτάσουμε στα, στο 2032, το, όπου έλυγε το σχέδιο του, το δασικό του 92. Παράλληλα, αυτή η επιφάνεια ε, καλύπτεται από ευκαλύπτους που φύονται όπως να είναι. Ε, είναι άγριοι ε, και είναι ένα ε, είδος Ε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ο ευκάλυπτος νίτενς, ο οποίος προσθέθηκε στα, φυτεμένα, στο φυτεμένο χώρο και πέρα από τον ευκάλυπτο globulus, ε, γιατί αντέχει πάρα πολύ στο κρύο. Ο ευκάλυπτος ε, νίτενς ε, θεωρείται από την Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου περιβάλλοντος της Ισπανίας ως ένα εξωτικό είδος, το οποίο επεκτείνεται, είναι χωροκατακτητικό, επικίνδυνο για τη βιοπικιλότητα και την λειτουργία των οικοσυστημάτων. αυξάνεται η... αυξάνονται οι ευκάλυπτοι και αυτό ευνοείται από ένα μοντέλο εκμετάλλευσης του δάσους ε, όλο και πιο έντονο ε, που, βασίζεται, που γίνεται για λόγους παραγωγής ξυλίας, ε, λόγω της μεγάλης προσθέμενης αξίας. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το γεγονός ότι οι μονοκαλλιέργειες πυρόφυλων ειδών οδηγούν σε όλο και περισσότερες πυρκαγιές, σε σε προβλήματα για την βιοπικιλότητα, σε ε, μόλυνση των ε, γεών, των ποταμόκολπων ε, με αγροχημικά προϊόντα και απορρίψεις κυταρίνης. Η βιοπικιλότητα μειώνεται καθώς προχωράει η διάβρωση λόγω των άμεσων οικονομικών απολειών και των αυξανόμενων κερδών από τις μονοκαλλιέργειες. Αυτό το δασικό μοντέλο συνεισφέρει στο να διασπαθήσουμε τεράστιες ποσότητες δημοσίων ε, ε, κονδυλίων μέσω του Πλάντιγα, ε, που είναι ένα σχέδιο καταπολέμησης της πυρκαγιάς και όπου κοστίζει κάθε χρόνο 150 εκατομμύρια ευρώ. καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν να ζητήσουν από την κυβέρνηση της Γαλλικίας να δημιουργήσει αμελητή ένα μορατόριο επαόριστο για τις νέες φυτεύσεις ειδών ευκαλύπτου σε όλη την επικράτεια της Γαλλικίας. Να απαγορεύσει την καλλιέργεια του ευκαλύπτους νήτες. Η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει μέτρα για την προοδευτική εκρίζωση αυτών των ειδών σε όλη την επικράτεια ε, και να δώσουμε σημαντική προστοχή ε, στις φυσικές περιοχές, στους φυσικούς χώρους, ε, στις γεωργικές γέες και στις γέες βοσκοτόπια. Να απαγορεύσουμε την αναδάσωση με όλα τα είδη του ευκαλύπτου ε, στη Γαλλικία. Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να κάνει τα απαραίτητα ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εμείς διαβάσαμε προσεκτικά τα γεγονότα που καταγγέλει ο αναφέρον. Ξέρουμε πάρα πολύ την κατάσταση που επικρατεί στη Γαλλικία. Σε ό,τι αφορά τα, τη χρήση κοινοτικών κονδυλίων, το, το πρόγραμμα για τη Γαλλικία του ΦΕΝΤΕΡ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014-2020, πρόβλεπε ε, την υλοποίηση του μέτρου 5.1 εξάντε για την αξιολόγηση του κινδύνου. Θα έπρεπε να γίνει είτε σε εθνικό επίπεδο ή σε περιφερειακό επίπεδο αξιολόγηση του κινδύνου λαμβάνοντα υπόψη την κλιματική αλλαγή. Αυτή η προϋπόθεση έχει ληφθεί υπόψη. Και γι' αυτό ακριβώς επειδή υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις έχουν εκταμιευθεί αυτό τα, αυτά τα κονδύλια. Ε, προβλέπονται 39,5 εκατομμύρια ε, ευρώ ε, από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής, ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης για την αντοχή μπροστά σε φυσικές καταστροφές κτλ. για τι επενδύσει και τη διαχείριση των καταστροφών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, για τις δασικέ πυρκαγιέ, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στηρίζει δράσεις όπω η εφαρμογή μοντέλων πρόληψη των κινδύνων με έγκαιρη ανείχνευση και εντοπισμό των κινδύνων, ε, με οχήματα, με μηχανήματα και εξοπλισμό για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και άλλων ειδών καταστροφών. Σας λέμε επίσης ότι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το πρόγραμμα ε, για τη Γαλλικία 2014-2020 ε, περιλαμβάνει επίσης μέτρα που ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ για να προλάβουμε πυρκαγιές βρασικού χαρακτήρα και τις ζημιές που προκαλούν αυτές, καθώς και φυσικές καταστροφές και, άλλα, και άλλων ειδών καταστροφές. Ε, επίσης, 16 εκατομμύρια ευρώ έχουν ε, προβλεφθεί εντός αυτού του προγράμματος για την αποκατάσταση των δασών. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο ευκάλυπτος αποκλείεται ρητά από αυτά τα είδη τα οποία μπορούμε να καλύψουμε στα πλαίσια της αναδάσωσης, της φυσικής αναδάσωσης. Δεν φυτεύουμε δηλαδή ευκάλυπτο. Σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη, όπως προτείνεται, του ευκάλυπτου στον κατάλογο των ευρωπαϊκών ειδών που είναι δυσδυτικά, χωροκατρακτητικά, η Κομισιόν δεν το θεωρεί αυτό πιθανό, δεν το θεωρεί δυνατό. Μια και το ψήφισμα υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2015 για το θέμα αυτό και αυτό το ψήφισμα μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από το ίδιο το Κοινοβούλιο. Επομένω, η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητε για να συμπεριλάβει σε ένα κατάλογο ευρωπαϊκού χαρακτήρα ένα είδο όπω τον ευκάλυπτο, που θεωρείται χωροκατακτητικό Μόνο η Επιστημονική Επιτροπή της Ισπανίας θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Με Ισπανούς επιστήμονες θα μπορούσε να αποφασίσει τη μεταχείριση που θα επιφυλάξει σε αυτό το είδος και θα δει αν το θεωρεί ε, χωροκατακτητικό είδος ή όχι. Yeah, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ε, να δώσω το λόγο στην κυρία Βαλίνα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ του να ρίχνουμε συνέχεια το φταίξιμο στις Βρυξέλλες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κακά που συμβαίνουν στη χώρα μας, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι σαφές ότι η κυβέρνηση της Γαλλικίας δεν έκανε το, μαθη... διάβασμά τη, δεν διάβασε, δεν έκανε τα μαθήματά της, δεν ήταν καλός μαθητής για να προλάβει τις δασικές πυρκαγιές. Και τώρα ζητάει χρηματοδότηση από την Ευρώπη για να κάνει επενδύσεις σε εξοπλισμό και σε απαραίτητο προσωπικό. Βλέπουμε τις καταστροφές που υφίσταται η Γαλλικία από τις πυρκαγιές. Και βλέπουμε επίσης πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση στην Αστούρια και τη Γαλλικία. Υπάρχουν αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τον τομέα της γεωργίας και τον τομέα της κτηνοτροφίας και του ζωικού κεφαλαίου. Άρα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει στις περιοχές αυτές στις οποίες αναφέρεται ο καταγγέλων. Διότι ε, καταλαβαίνετε ότι όντως ε, χάνονται διάφορε θέσει απασχόληση όταν καταστρέφονται γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε όλε αυτέ τι περιοχέ. Αυτό δείχνει ότι όταν υπάρχουν ε, γεωργοί, όταν υπάρχουν ζώα τα οποία βόσκουν και καθαρίζουν τα δάση, δεν προχωρούν οι φωτιές. Στην ε, Γαλλικία όμως και στην ε, Αστούρια παρατάμε και εγκαταλείπουμε τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, εγκαταλείπουμε τις γέες και χρειαζόμαστε δημόσιο χρήμα μετά για να διορθώσουμε τα λάθη. Η Κομισιόν σε ένα ανακοινωθέν τύπου ε, τον περασμένο Σεπτέμβριο αναγνώρισε ότι η φύτευση ε, ειδών στα δάση προωθούν τις πυρκαγιές και επιτρέπουν την εξάπλωσή τους. Επίσης ε, υπάρχει αυτή η μονοκαλλιέργεια του ευκάλυπτου στην ε, Ισπανία. Ακριβώς κάνει το αντίθετο από αυτό που θέλουμε για να καταπολεμήσουμε και την κλιματική αλλαγή κατά την απόψή μας και για να δώσουμε περισσότερες δυνατότητε στις τοπικές οικονομίες, θα πρέπει να έχουμε κοινέ στρατηγικές σε όλες ε, τις ε, κοινότητες και δήμου για να ελκύσουμε πληθυσμό, για να έχουμε παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες και να έχουμε μια πολιτική υπέρ των δασών και, κατά της πρόληψης... και υπέρ της πρόληψης των πυρκαγιών. Πιστεύουμε ότι αυτή η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Θα πρέπει να στείλουμε μία επιστολή στις γαλλικιανές αρχές για να εξηγήσουμε ότι πρέπει να μας δώσουν στοιχεία για το πώς ξόδεψαν κάθε ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ε, στην Αστούρια που είναι η περιοχή μου και εμείς λάβαμε κονδύλια και δυστυχώς τα ξοδέψαμε ε, κακήν κακό, τα ξοδέψαμε λάθος και πρέπει να τα επιστρέψουμε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν πάντα πρέπει να ερευνούμε πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια. Ε, χάρη στην έρευνα που έγινε, ε, αποδείχθηκε ότι υπήρχε κακοδιαχείριση αυτών των κονδυλίων και η Αστούρια, η περιοχή μου δηλαδή, έπρεπε να επιτρέψει αυτά τα κονδύλια. Επίση, νομίζω θα πρέπει να κάνουμε μια μελέτη για τι ζώνε όπω η Γαλλικία, η Αστούρια και όλη η ακτή, όπου είχαμε μεγάλη απώλεια πληθυσμού, για να καταλάβουμε ακριβώς τι κάνουμε με τα λεφτά της Ευρώπης και να δούμε τι εναλλακτικέ έχουμε. Μετά από τόσα χρόνια, ίσω πρέπει να σκεφτούμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν, κάνει, δεν πετυχαίνει αυτό που θα έπρεπε. Θα πρέπει να κάνουμε μια μελέτη αντικτύπου για να δούμε η ΚΑΠ τι επίπτωση είχε στι διάφορε χώρε. Γιατί αν υπάρχει αποψήλωση ή εγκατάλειψη του πληθυσμού κτλ. σε κάποιε περιοχέ, τότε ε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε μήπως αυτά τα προβλήματα, ας πούμε, η μείωση του πληθυσμού προκαλούνται από την κοινή γεωργική πολιτική. Ε, gracias, Η επόμενη συνάδελφος, η κυρία Σέρα Ροδρίγεθ. Καταρχάς, μιλάμε για κακή χρήση, από ό,τι είπε ο αναφέρον που φέρνει αυτό το θέμα ενώπιόν μας, ενώπιον της Επιτροπής. Μιλάμε λοιπόν για χρήση και κακή χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων. σε ό,τι αφορά την πρόληψη ε, και την κατάσβεση πυρκαγιών στην Καλικία. Θα πρέπει να δούμε πού πήγε αυτό το χρήμα. Πρώτον. Επίση, θα πρέπει να δούμε αν λαμβάνονται σωστά μέτρα για να υλοποιηθούν οι στόχοι. Όπω επίση μα είπε η Κομισιόν, τι μα λέει, ότι τα χρήματα αυτά από τα ταμεία θα πρέπει να δοθούν για μέτρα κατά καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής. Και θα πρέπει οι προτάσεις αυτές να είναι ουσιαστικές για την αντίσταση στην κλιματική αλλαγή. Θα, τώρα, με το να επιτρέπουμε τις φυτεύσεις ευκάλυπτο ή ε, με την μονοκαλλιέργεια του ευκαλύπτου, είναι σαν να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Η Κομισιόν, όπως είπε και η συντροφός μου, αναγνώρισε ότι ένα από τα προβλήματα βρίσκεται στο γεγονός ότι υπάρχει γίνονται πυρκαγιές και φουντώνουν οι πυρκαγιές λόγω των πυρόφιλων ε, ειδών που έχουμε. Και ο ευκάλυπτος είναι τέτοιο πυρόφιλο είδος. Ε, σε ό,τι αφορά το ΦΕΑΔΕΡ και το πρόγραμμα 2014-2020 ε, για τη Γαλλικία. Τον Αύγουστο του 2018 δώσαμε 2.000 ευρώ δημόσιο χρήμα για 16 μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ε, τις πω, πώς. Ε, αντικαθιστώντας τα, τους ευκάλυπτους με πλατήφυλλα ε, δέντρα στα δάση ή αυτόχθονα άλλα είδη. Κοιτάξτε αυτή τη φωτογραφία, Κομισιόν, που είναι από μια επίσκεψη που κάναμε, μια σύντροφος και εγώ, σε ένα δάσος ε, με αυτόχθονα είδη, το οποίο κόψαμε όμως για να φυτέψουμε ευκαλύπτους. Κάτι που απαγορεύει η νομοθεσία. Και όμως έγινε. Και μάλιστα έγινε σε δασική περιοχή, όπου η κυβέρνηση της Γαλλικίας με, ε, με το δασικό σχεδιασμό που κάνει λέει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ευκάλυπτος κανονικά. Και αυτό γίνεται τη στιγμή που το ξέρουν οι αρχές. Το ξέρουν οι αρχές και γίνεται παρόλα αυτά. Θα ήθελα η Κομισιόν να ερευνήσει αυτή την κατάσταση και τη χρήση αυτών των δύο εκατομμυρίων που υποτίθεται θα δινόταν για να αντικατασταθεί ο ευκάλυπτος από αυτόχθονα είδη. Επίσης έγινε λόγο για την εγκατάλειψη του περιβάλλοντος. Είναι προφανές αυτό. Δεν χρειάζεται να μπω σε περισσότερε λεπτομέρειε. Η Άγχελα, η, ε, συνάδελφο, μου, μίλησε αρκετά. Ποια είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που λείπουν. Γιατί στη Γαλλικία παράγεται, μάλλον ε, προκαλούνται το 70% των πυρκαγιών σε όλη την Ισπανία και καίγεται το 56% των δασών ε, που καίγονται γενικά σε όλη την Ισπανία. Το 56% ανήκουν στην Γαλλικία. Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί καίγονται πολύ περισσότερες επιφάνειες στη Γαλλικία από, από αλλού. Θα πρέπει να έχουμε ένα δασικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στον ευκάλυπτο. Αυτό, αν το λέμε, είναι σαν να λέμε ότι επίτηδες δεν θα υλοποιήσουμε τους στόχους ε, καταπολέμησης της ε, κλιματικής αλλαγής. Το δημόσιο χρήμα, τα λεφτά των φορολογουμένων, των Ευρωπαίων φορολογουμένων δεν χρησιμοποιούνται σωστά λοιπόν, εάν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το μοντέλο ας πούμε, για τα δάση. Επίσης, το να δίνουμε σε ιδιωτικές εταιρείες το καθήκον της πυρόσβεσης, αυτό είναι πολύ πιο ακριβό από το να προσλάμβανε δημοσίου υπαλλήλου η δημόσια διοίκηση για το καθήκον αυτό, για την πυρόσβεση. Αυτό θα πρέπει να το ελέγξουμε. Αν έχει νόημα δηλαδή να αναθέτουμε αυτό το έργο σε ιδιωτικέ εταιρείε. Το δημόσιο χρήμα που χρησιμοποιείται για την πρόληψη και την ε, πυρόσβεση οδηγεί ουσιαστικά σε επισφαλείς ε, συνθήκες εργασίας για το προσωπικό το οποίο κάνει αυτή την ε, πυρόσβεση. Κι όμως, αυτό που θα πρέπει να μας είναι πώς θα αποφύγουμε αυτές τις, ε, αυτά τα προβλήματα, δηλαδή το να βάζουμε τους εργαζομένους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Τέλος. Υπάρχει το Εθνικό Δικαστήριο το οποίο ερευνά διάφορα θέματα ε, για την καθαρότητα του αέρα. Ε, και επίσης ε, γίνεται μια έρευνα για το πώς δίδονται τα δημόσια έργα, πώς κατανέμονται στην, στην Ισπανία γενικά. Στην Ισπανία δεν έχουμε μέτρα ανθεκτικότητας, δεν υπάρχει σοβαρή πρόληψη θα πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερες ε, πληροφορίες από τις αρχές της Γαλλικίας. Και μάλιστα θα έλεγα η Επιτροπή να κάνει μία επίσκεψη στο μέλλον για να δούμε επιτόπου τι συμβαίνει με τις πυρκαγιές, τι γίνεται με το δασικό μοντέλο και τι γίνεται με την εγκατάλειψη στη μοίρα του του περιβάλλοντος. Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μιλαμών. Μετά από αυτά που άκουσα, και επειδή θέλω να σεβαστώ τους προλαλήσαντες, ε, θέλω να πω ότι σέβομαι τα άτομα που μίλησαν, δεν δε σέβομαι τις απόψεις τους, γιατί ε, είναι σαν κασάνδρες. Ε, παρουσιάζουν μια ζωφερή εικόνα. Υπάρχει και μια άλλη εικόνα για τη Γαλλικία. Δεν συμφωνώ με αυτά που λένε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι έγινε ανάλυση κινδύνου. Έγινε από την κυβέρνηση της ε, Γαλλικίας, υπάρχουν ε, σχέδια πρόληψης, ε, κατεπήγοντος, υπάρχει το σχέδιο Πλαντίγκα. Η Κομισιόν μας εξήγησε τι προσπάθειες έκανε η τοπική κυβέρνηση και τι, πώς εξοδεύτηκαν τα λεφτά από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Καταρχάς πρέπει να δούμε τα γεγονότα, τα στοιχεία. Το 2014-2018 η Γαλλικία ε, είχε 2.300 πυρκαγιές ετήσιες. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο, αλλά σε σχέση με προηγούμενα έτη είχαμε ε, μείωση κατά 50% των πυρκαγιών, όπου είχαμε πάνω από 3.500 ε, πυρκαγιές. Συγγνώμη, 230 πυρκαγιές, όχι 2.300. Μιλάω για ετήσια νούμερα, έτσι. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα στο, στις δασικές γέες ε, στη Γαλλική. Είναι διαφθορτικό πρόβλημα. Επίσης το γεγονός ότι τα δάση βρίσκονται στα χέρια διωτών, ότι υπάρχουν, ε, ο πληθυσμό μειώνεται, δεν υπάρχει σωστή διαχείριση, ότι πολλοί γεωργοί έχουν εγκαταλείψει ε, τις γέες τους. Από τη δεκαετία του 50 ας πούμε, μέχρι σήμερα έχουν φύγει ε, τη δεκαετία του 50 είχαμε πάνω από 500.000 γεωργού στη Γαλλική... και τώρα έχουμε 46.000. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο μειώθηκε ο πληθυσμό. Τώρα υπάρχει αυτή η βούληση να εξασφαλιστεί η οικονομική δραστηριότητα, να βελτιώθει η πρόληψη των πυρκαγιών ε, και να αποκατασταθεί η γεωργική δραστηριότητα. Ε, μία βιώσιμη διαχείριση επίσης των βουνών δεν είναι τίποτα το απαρχαιωμένο ε, σε όλα αυτά που σας είπα. Όπως λέει ο αναφέροντας, πέρυσι ε, αναθεωρήθηκε το πλάνο αυτό το δασικό του 1992, θα τα ξέρει το κοινό. Είναι δημόσιες πληροφορίες και τώρα ε, είναι ανοιχτό να το διαβουλευτεί οποιοδήποτε πολίτης. Επίσης υπάρχει υπάρχουν μεταρρυθμίσεις. Ε, μην μένουμε με αυτή την ε, εικόνα του, της δεκαετίας του 90. Έχουν ε, γίνει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Επίσης, μία επιτροπή από διάφορα κόμματα ε, υιοθέτησαν κάτι, κάποια συμπεράσματα ε, με, τους, με το Λαϊκό Κόμμα και με τους σοσιαλιστές της Γαλλικίας. Δημιουργήθηκε μάλιστα και μία ομάδα εργασία με πυρογνώμονε κτλ. για να δουν πώ μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο επώδυνο θέμα και σημαντικό. Τι γίνεται με τις ε, πυρκαγιές λόγω των ευκαλύπτων κτλ. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν κάποιοι, κάποια άτομα που εκ προθέσεως καίνε τα δάση. Ε, το 75% των ε, πυρκαγιών, ε, των 2.300 τελικά πυρκαγιών, το 75% τα 2 τρίτα δηλαδή, ε, είναι εμπρισμοί, είναι πυρκαγιές Ε, 10 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020 για να εξυγχρονίσουμε τα οχήματα πυρόσβεση. Από το ΦΕΑΝΤΕΡ, το Γεωργικό Ταμείο, δηλαδή για την άπτυξη της υπαίθρου, Έχουμε δώσει 120 εκατομμύρια για την πρόληψη και τη βοήθεια για, τις, για αυτούς που έχουν υποστεί ε, φυσικές καταστροφές. Από το Γεωργικό Ταμείο, έτσι. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τα ταμεία και, το, και τα δύο γεωργικά ταμεία και το Ταμείο Εγγύσεων και το Ταμείο για την Ανάπτυξη Πέθρου. Άρα χρησιμοποιούνται σωστά τα κονδύλια. Τώρα για το να ταξινομηθεί ο ευκάλυπτος ως χωροκατακτικό είδος, καταρχάς υπάρχει μια ευρωπαϊκή διαδικασία γι' αυτό. Στην Ισπανία ούτε καμία άλλη χώρα δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ε, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχει κανένα κατάλογο, το λέω αυτό στον αναφέροντα. Δεν υπάρχουν κατάλογοι σε αυτό το ψήφισμα. Τρίτον, αυτή η έκθεση της ε, Επιστημονικής Επιτροπής του 2017. Δύο μήνες μετά, το Υπουργείο Γεωργίας ε, είπε ότι αυτή η έκθεση είναι άκυρη. Είπαν ότι είναι λάθος αυτά που λέει η έκθεση. Ότι δεν είναι σωστά αυτά που λέει για, την, για τον ευκάλυπτο ως χωροκατακτητικό είδος. Υπάρχει απλώς ένας ε, δήμαρχος ο οποίος λέει ότι είναι χωροκρατικό ύφος, αλλά η κυβέρνηση της Ισπανίας διαφωνεί Ούτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούμε ότι είναι χωροκρατικό είδο ο ευκάλυπτο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλάμε μόνο, παντά, μόνο πλευρά, α πούμε. Πρέπει να δούμε όλη την ε, ε, φωτογραφία. Από τα δάση τα οποία κάηκαν, ε, μόνο το 7,5% καλύπτονταν από ευκάλυπτους. Από ευκαλύπτους. Ε, τι να σας πω. Ε, με βάση τα δεδομένα, δηλαδή, έχει λιγότερε πυρκαγιέ εκεί που έχουμε ευκαλύπτου. Με βάση τα δεδομένα που έχω, έτσι. Ε, και τελειώνω, Πρόεδρε. Εμεί στη Γαλλικία Θέλουμε να έχουμε δάση ε, με βιοπικιλότητα. Αλλά δεν θα πρέπει να τιμωρούμε κάποια είδη, δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι κάποια είδη είναι κακά και προβληματικά. Απλώ να τα ελέγχουμε. Θα πρέπει να ελέγξουμε την επέκταση του ευκαλύπτου, αλλά δεν θα πρέπει να απαγορεύσουμε την φύτευσή του. Ε, πέρα από τα κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη που μπορεί να μας δώσει. Έτσι. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, η κυβέρνηση Γαλλικίας δεν επιδότησε την ε, φύτευση του ευκαλύπτου. Ε, επιδότησε αντίθετα τη φύτευση της καστανιάς, αλλά όχι του ευκαλύπτου. Έχουμε πάνω από 450.000 εκτάρια με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τη Γαλλικία, δεν είναι αυτά τα νούμερα σωστά. 250.000 εκτάρια είναι αυτά που καλύπτονται από ευκαλύπτου, όχι 350.000. Δεν ξέρω αν είναι πόλεμο με τα νούμερα τώρα, αλλά τι να σα πω, το να αφήσουμε την ε, αναφορά αυτή ανοιχτή και να ζητάμε περισσότερε πληροφορίε ή να χαρακτηρίσουμε, εν πάση περιπτώσει, τον ευκάλυπτο χώρο κατακτητικό είδο τη στιγμή που δεν συμφωνεί η κυβέρνηση τη Ισπανία. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν έχει πολύ νόημα δηλαδή αυτή η συζήτηση. Έχουμε κάποιες ε, ιδέες ε, που υποστηρίζουμε μανιακά, ας πούμε, κατά του ευκαλύτου. Δεν είναι σωστά αυτά τα νούμερα και αυτά τα στοιχεία. Ρόζα Εστερά Φάργκουτ. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Πάκο. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς του αναφέροντες. Θέλω να σας πω ότι τα δύο θέματα με τα οποία ασχολείται η αναφορά σα καταρχάς την πιθανή κακοδιαχείριση των χρημάτων του ΦΕΑΝΤΕΡ. Δεν συμφωνώ με αυτήν. Η Κομισιόν ε, εξετάζει πολύ λεπτομερώς την, ε, τον τρόπο που δαπανώνται αυτά τα κονδύλια. Ε, ο έλεγχος είναι πάρα πολύ λεπτομερής. Υπάρχει θέμα διαφάνειας, θέμα, θα υπήρχε θέμα διαφάνειας, θα υπήρχε θέμα ασφάλειας δικαίου αν δεν γινόταν αυτό, αν δεν γινόταν σοβαρή έλεγχη. Υπάρχουν σχέδια που μπορεί να σας φαίνονται ε, άσχημα ή καλά. Το βασικό είναι ότι είναι νόμιμα. Όπω είπε και η Κομισιόν, υπάρχει απόλυτη νομιμότητα. Τα κονδύλια των γεωργικών ταμείων ε, ασχολούνται για πρόληψη, για εκρίζωση χωροκατακτητικών ειδών. Ε, μιλάμε για πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει μια πολύ λεπτομερή έκθεση ε, για τα δύο γεωργικά ταμεία ε, και πώς εξοδεύονται αυτά τα κονδύλια για τον εξυγχρονισμό των ε, οχημάτων. Αντικαθιστούμε το 50% των οχημάτων για την πυρόσβεση. Όλα αυτά έγιναν για να μειωθούν οι πυρκαγιές και έχουν μειωθεί κατά 50%. Σημαντικό νούμερο και για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το οικοσύστημα. Πέρα από τη μείωση των ε, δασικών πυρκαγιών, μην ξεχνάτε ότι και ένα μεγάλο τμήμα αυτών των ε, πυρκαγιών είναι εμπρισμοί. Και πολύ λιγότερε πυρκαγιέ είναι από πραγματικά φυσικά αίτια. Επομένω, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ζητήσουμε τίποτα από τα ταμεία. Ούτω ή άλλω, η διάγνωση τη Κομισιόν είναι ότι υπάρχει απόλυτα σωστά χρήση των κονδυλί... σωστή χρήση των κονδυλίων με απόλυτη νομιμότητα. Η ταξινόμηση τώρα του ευκάλυπτου ω ε, χωροκατακτητικού είδου δεν είναι αρμοδιότητα τη Γαλλικία. Ούτως ή άλλως, κανένας δεν ε, δίνει επιδοτήσεις για να φυτέψουμε ευκάλυπτο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Παρότι το έχει ζητήσει μια επιστημονική επιτροπή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ε, το Υπουργείο Γεωργίας δεν το δέχτηκε. Και, εν πάση περιπτώσει, ποιο αποφασίζει για κάτι τέτοιο, το Κοινοβούλιο, με αυτόνομο τρόπο. Εδώ, παραδείγματο χάρη, εδώ που είμαστε 28 χώρε, το συζητήσαμε το θέμα και, και είπαμε είναι ή δεν είναι. Και αποφασίσαμε ε, με τα λόγου γνώση ότι δεν είναι χωροτακτητικό είδο. Βεβαίω είναι ένα είδο το οποίο θα πρέπει να ελέγχεται. Έχει παρόλα αυτά παραγωγική αξία. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Επομένως, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν συμφωνώ με τα προβλήματα που αναφέρει η έκθεση αυτή, δεν υπάρχει πρόβλημα με τον ευκάλυπτο. Και ούτω ή άλλω ο κατάλογο αυτό για τα χωροκρατητικά είδη ε, έχει κλείσει από πλευρά Κοινοβουλίου από το 2015. Το βασικό είναι ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα, υπάρχει απόλυτη νομιμότητα και υπερασπιζόμαστε την νομιμότητα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα διάφορες παρεμβάσεις. Στηρίζω τους συντρόφους και τις συντρόφισσες. Υπάρχει πρόβλημα συνέπειας, όπως βλέπουμε, γιατί η βασική λέξη, λέξη κλειδί είναι η συνέπεια. Από τη μία, ζητάμε σχέδια πρόληψης και πυρόσβεσης και λέμε ότι είμαστε οι καλύτεροι πρωταγωνιστές στον αγώνα της, ε, κατά της κλιματικής αλλαγής. Και από την άλλη, το να εμένουμε σε ένα μοντέλο το οποίο είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό, δηλαδή που είναι η μονοκαλλιέργεια ευκάλυπτου, αυτό είναι, είναι πλήρης ασυνέπεια. Κάναμε δύο συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα το να μας λέτε ότι είμαστε ζωφεροί, ας πούμε, ότι φέρνουμε την καταστροφή, καταστροφολόγοι κτλ. είναι σαν να μην έχετε ε, συνέστηση και να μην καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Α είμαστε λιγάκι προσεκτικοί, έτσι. Γιατί Ισπανία, Γαλλικία, Ανδαλουσία, Πορτογαλία είναι περιοχές και χώρες που επλήγησαν πάρα πολύ από τις πυρκαγιές. Βλέπετε ότι έχουμε τόσο διαφορετικές απόψεις. Δεν υπάρχει συνέπεια. Να μην ξεχνάμε ότι οι συνέπειες της πολιτικής είναι σημαντικό πράγμα στην Ευρώπη και αυτό θα πρέπει να μην ξεχνάμε. Δεν θα πρέπει δηλαδή από τη μία να επιδοτούμε και από την άλλη να ξεκάνουμε αυτό που επιδοτούμε. Δεν είναι σοβαρό αυτό. Ας κάνουμε λοιπόν κάτι που μου φαίνεται εμένα συνεπές και λογικό. Ας κάνουμε μια επίσκεψη, πάμε στην ε, Γαλλικία από διάφορες πολιτικές ομάδες για να δούμε αυτά τα νούμερα, τα οποία λένε ορισμένοι ας πούμε, για να δούμε αν όλα αυτά που μας λένε οι μεν και οι δεν είναι σωστά. Α πάμε επί τόπου, όλοι μαζί. Το έχουμε ξανακάνει αυτό. Γιατί να μην το κάνουμε και στη Γαλλική να δούμε την πραγματικότητα, να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα με το μοντέλο, να συζητήσουμε αυτό το μοντέλο και να το συζητήσουμε δημοκρατικά. Να μην κλείσουμε λοιπόν την αναφορά. Σα ευχαριστώ που την παρουσιάσατε. Να πάμε επί τόπου με μια επίσκεψη, να δούμε τέλο πάντων τι συνέβη εκεί. Σα ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Θα πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πήραν το λόγο. Και άκουσα να προτείνονται δύο λύσεις. Η μία είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Η δεύτερη πρόταση ήταν να κλείσει η αναφορά ή μάλλον να σταλεί επιστολή στις αρχές της Γαλλικίας για να ε, γνωρίζουν το πρόβλημα. Περνάμε στην ψηφοφορία. Μόνο οι παρόντε ευρωβουλευτέ έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Ε, Ποιο είναι υπέρ του να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Τρει. You were influenced, but, but uh, Η δεύτερη δυνατότητα είναι να στείλουμε επιστολή στις αρχές της Γαλλικίας και να κλείσουμε την αναφορά. Ποιος είναι υπέρ αυτής της λύσης. Πρόβλημα διαδικαστικό. Κανονικά κλείνει ο αναφέροντας, έτσι. Πριν αποφασίσουμε θα κάνουμε την ε, αναφορά, πρέπει να του ξαναδώσουμε το λόγο. Uh, who in close Ποιος είναι υπέρ του να κλείσει η αναφορά. Η πλειοψηφία. Κύριε Λόπες Πέρες, θα κλείσει η αναφορά. Έχετε φυσικά το δικαίωμα. Να συνεχίσετε να παρακολουθείτε το θέμα αυτό στο μέλλον. Έχει ληφθεί η απόφαση, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Το πρόβλημα του ευκαλύπτου ε, προάγεται αυ... λόγω του τρόπου που εκμεταλλευόμαστε τα βουνά. Δεν έχει προστιθέμενη αξία. Η δασική πολιτική της κυβέρνησης της Γαλλικίας είναι να προωθήσει τη φύτευση ευκαλύπτων. βλέπετε ότι η κυβέρνηση της Γαλλικίας στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί δημόσιο χρήμα και το δίνει σε στην εταιρεία η οποία φυτεύει ευκολύπτους. Δεν μπορούμε να ξοδεύουμε τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ε, η διαχείριση των βουνών είναι προβληματική. Πρέπει να ξαναδούμε το μοντέλο αυτό. Για μένα λοιπόν η αναφορά αυτή πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Σα ευχαριστούμε πολύ. E, Όπω ξέρετε, έχουν ήδη αποφανθεί όμω οι ευρωβουλευτέ για την αφορά αυτή. Λοιπόν, α ακούσουμε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν στην Επιτροπή μας τον καθηγητή Μισελ Φορ ε, από τα Πανεπιστήμια Μάστρεκτ και Ρότερνταμ. Κύριε καθηγητά, καλώς ήλθατε στην Επιτροπή μας. Έχετε 15 λεπτά για να κάνετε την παρουσίαση της πολύ ενδιαφέρουσα αυτής μελέτης. Ένα τεχνικό θέμα δεν είναι. Ε, διαδικαστικό, έτσι, θέλω να θέσω. Ψηφίσαν τα διάφορα κόμματα. Αλλά υπάρχει μια πολιτική ομάδα εδώ η οποία κατέβηκε μαζικά και εμποδίζει την πραγματική δημοκρατία. Κλείνει δηλαδή η αναφορά γιατί κατέβηκε μαζικά μια πολιτική ομάδα, ένα κόμμα. Γι' αυτό έκλεισε η αναφορά. Αλλιώ δεν θα κλείνε. Τελείωσε. Έκλεισε η συζήτηση εδώ πέρα. Όσοι είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν, ψηφίσανε, λέει ο πρόεδρο. Είχατε τέσσερι ψήφου εσεί. Έχει κλείσει η συζήτηση. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσω την μελέτη μας αυτήν. Βρίσκομαι εδώ μαζί με την κυρία Κέντζη, την δόκτωρα Κέντζη, και έχουμε από κοινού συντάξει τη μελέτη αυτή που έχετε ενώπιόν σας. Και βρισκόμαστε εδώ διότι έχουν εκφραστεί αρκετές ανησυχίες στις διάφορες αναφορές που επεξεργάζεστε. Έχουμε εκπονήσει λοιπόν μια μελέτη 140 σελίδων και στα 15 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου δεν πρόκειται να σας παρουσιάσω και τις 140 αυτές σελίδες. Θα ήθελα απλώς να τονίσω κάποιες πτυχές της μελέτης αυτής. Καταρχά, προσπαθήσαμε να δούμε ποιε είναι οι βασικέ ανησυχίε που εκφράζονται μέσω των αναφορών αυτών. Είδαμε ότι πολλοί αναφέρονται, αναφέρονται στο ζήτημα τη πυρηνική ασφάλεια και ιδίω τη διασυνοριακή πυρηνική ασφάλεια, με το τιονς 2 για παράδειγμα. Επίση, άλλε αναφορέ ζητούν να κλείσουν κάποια πυρηνικά εργοστάσια, κάποια πυρηνική σταθμή. Γενικέ απαιτήσει αυτέ θα έλεγα περισσότερο. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι υπάρχουν μεγάλε διαφορέ ανάμεσα στα συστήματα ευθύνη από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και υπάρχουν άλλοι αναφέροντες που ζητούν ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα ανάληψης ευθύνης και ασφάλισης αστικής ευθύνης. Πάνω στα ζητήματα λοιπόν αυτά βασίσαμε τη μελέτη μας κύριε Πρόεδρε, πάνω στις βασικές αυτές ανησυχίες οι οποίες εκφράζονται με μεγάλη σαφήνεια και οι οποίες ε, οι περισσότερες αναφέρονται στο ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια όσον αφορά τα συστήματα ανάληψης ευθύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς συμφωνούμε με την άποψη αυτή και θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, ποιο είναι το γενικότερο νομικό πλαίσιο όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται πάρα πολύ στο διεθνές πλαίσιο. Εδώ έχουμε την σύμβαση CNS για την πυρηνική ασφάλεια του 1994 που βασίζεται σε πρότυπα τα οποία προκύπτουν από το Διεθνή Οργανισμό Τοπικής Ενέργειας. Αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό, κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε διατάξεις ε, ήπιου δικαίου, μη δεσμευτικέ ουσιαστικά διατάξει. Και έπειτα έχουμε και κάποιε διατάξει πρότυπα που προκύπτουν από την Υπηρεσία Πυρηνική Ενέργεια του ΟΣΑ. Στο δεξί τμήμα της διαφάνειας βλέπετε, αν θέλετε, τα ευρωπαϊκά μέσα. Καταρχάς, τη συνθήκη Ευρατόμ. Τι κάνει η συνθήκη ευρατόμ; Ευρατόμ, θέτει κάποια βασικά πρότυπα. Αλλά και πάλι η συνθήκη Ευρατόμ εστιάζεται περισσότερο στην προστασία των εργαζομένων και του κοινού και όχι τόσο πολύ στο ζήτημα της πυρηνικής ασφάλειας αυτής καθεαυτής. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε και μία οδηγία βασικών προτύπων. Την έχουμε την οδηγία αυτή, αλλά και αυτή βασίζεται ιδιαίτερα, επικεντρώνεται μάλλον περισσότερο στην ακτινοβολία, τη ραδιενέργεια και λέει ότι θα πρέπει τα επίπεδα της ραδιενέργειας αυτά να είναι στο δυνατόν, όσο δυνατόν πιο εφικτό, πιο χαμηλά. Και έπειτα έχουμε και την οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια, μια άλλη κοινοτική οδηγία, η οποία είναι ενισχύει. Βλέπετε λοιπόν ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο βασίζεται πάρα πολύ στο διεθνές soft law, στο διεθνές ήπιο δίκαιο και στα σχετικά πρότυπα τα οποία έχουμε από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ή από τη Σύμβαση για την Πυρηνική ε, Ασφάλεια και τα πρότυπα αυτά του soft law γίνονται δεσμευτικά μόνο και μόνο επειδή έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών μέσω των κοινοτικών οδηγιών. Παρ' όλα αυτά, τα μοντέλα πυρηνική ασφάλεια και τα πρότυπα πυρηνική ασφάλεια που ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αρκετά ασθενή. Εξαρτώμεθα πάρα πολύ από τόσα προβλέπεται στα πλαίσια τη εθνική νομοθεσία, από τόσα κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο βλέπουμε επίσης στη μελέτη αυτή, κύριε Πρόεδρε, είναι το τι ισχύει όσον αφορά την διασυνοριακή διαχείριση του πυρηνικού κινδύνου. Έχουμε και εδώ διάφορα εργαλεία. Ορισμένα από αυτά είναι εξαιρετικά και έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την ετοιμότητα και την ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε επίσης και το σύστημα IQRI, το σύστημα ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες και αυτό το οποίο βλέπετε ουσιαστικά είναι ότι υπάρχει ένα ευρύ καθεστώ διαφορετικών προτύπων και διαφορετικών διατάξεων, ακόμα και τη διαχείριση αυτή τη διαστοριακή του πυρηνικού κινδύνου. Πάλι, αν με ρωτήσετε τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα σα έλεγα ότι ελάχιστα είναι τα ευρωπαϊκά δεσμευτικά όργανα τα οποία διαθέτουμε. Και ένα ανάλογο μοντέλο έχουμε κύριε Πρόεδρε, αν δείτε τα συστήματα ασφάλειας και ευθύνης που ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ουσιαστικά τι έχουμε. Συστήματα ευθύνη και ασφάλιση, τα οποία πορέουν κυρίω από, την... από το Διεθνή Οργανισμό Ατομική Ενέργεια, καθώ επίση και από την Υπηρεσία Πυρηνική Ενέργεια του ΟΣΑ. Βλέπετε ουσιαστικά ότι ό,τι ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάλι απορρέει από τις διεθνείς συμβάσεις. Δεν έχει εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο καμία ξεχωριστή νομοθεσία όσον αφορά την πυρηνική ευθύνη και ασφάλεια. Α μην ξεχνάμε ότι όταν ξεκινήσαμε το 1960 με τη χρησιμοποίηση πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια, είχαμε τι συμβάσει ε, τη λεγόμενη πρώτη γενιά. Έχουμε καταρχάς την Συνθήκη των Παρισίων του 1960, τη Συνθήκη των Βρυξελών του 1963 και έπειτα και την Σύμβαση της Βιέννης του 1963 πάνω στην οποία βασίζεται ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια κάποια πολυπλοκότητα γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο ένα καθεστώς, αλλά πάλι που συμμετέχουν σε άλλο. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Και κυρίε και κύριοι, ε, μια πιο έντονη δραστηριότητα ξεκίνησε μετά το ατύχημα του Τσερνομπίλ, το οποίο αποτέλεσε αφύπνιση για τη διεθνή κοινότητα, η οποία τότε συνειδητοποίησε ότι οι διεθνείς συμβάσεις με την τότε μορφή του σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να παράσχουν την επαρκή αποζημίωση που απαιτείται. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε διεθνείς συμβάσεις δεύτερης γενιάς. Βλέπετε τη διαφάνεια αυτή, η οποία φαίνεται να είναι αρκετά εντυπωσιακή. Εμφανίζονται εδώ πέρα πέντε διαφορετικά εργαλεία μετά το ατύχημα του Τσερνομπίλ. Βλέπετε εδώ πέρα το κοινό πρωτόκολλο του 1988 και διάφορα πρωτόκολλα τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν τη Σύμβαση των Παρισίων, τη Σύμβαση της Βιέννης και τη Σύμβαση των Βρυξελών. Αλλά το Τσερνομπίλ έλαβε χώρα, κύριε Πρόεδρε, πριν από 30 χρόνια και πάνω από 30 χρόνια και βλέπετε ότι δύο από τις συμβάσεις αυτές ακόμα δεν έχουν τεθεί σε ισχύ. Και κατά την απίνη μας γνώμη θεωρούμε ότι ακόμα και οι ε, προσαρμογές αυτές που δεν έχουν τεθεί σε ισχύ ήδη έχουν απαρχαιωθεί. Επομένως κάτι πρέπει να κάνουμε επιγόντως. Ας δούμε τώρα ποιος πληρώνει και τι ακριβώς σε περίπτωση ατυχήματος. Τα έχουμε συνοψίσει όλα αυτά στη διαφάνεια που έχετε ενώπιόν σα. Βλέπετε εδώ πέρα ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε εκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε λοιπόν ότι βάσει συγκεκριμένων συμβάσεων όπω η Σύμβαση των Παρισίων προβλέπεται ότι ο οικονομικό φορέα που διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό σύμφωνα με τι συμβάσει τη πρώτη γενιά πρέπει να καταβάλει 57 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, οι συμβάσει αυτέ θα πρέπει να περάσουν στο εθνικό δίκαιο και τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέψουν και ανώτερα ποσά βλέπετε ότι στι συμβάσει τη πρώτη γενιά δεν έχουμε μόνο τον οικονομικό φορέα του πυρηνικού σταθμού, αλλά έχουμε επίση ω υπεύθυνο και το κράτος εγκατάσταση, το οποίο καλείται και αυτό να καταβάλει μια αποζημίωση. Αν συγκρίνετε τα ποσά, συνειδητοποιείτε τελικά ότι ο οικονομικό φορέα πληρώνει πολύ λιγότερα σε αποζημίωση από ότι ο κρατικό φορέα, από ότι οι κρατικέ αρχέ. Ουσιαστικά εδώ πέρα όλα αυτά παίρνουν τη μορφή μια επιδότηση τη πυρηνικής ενέργεια. Θα μπορούσε κάποιο να πει, πολύ ωραία, τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν με τις συμβάσεις της δεύτερης γενιάς. Και αυτό ισχύει εν μέρη διότι βλέπουμε ότι καθίσταται πιο υπεύθυνο αυτή τη φορά ο Οικονομικός Φορέας λειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου. Καλείται, όπως βλέπουμε τώρα, να πληρώσει 500 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αλλά έρχεται έπειτα και το κράτος εγκατάσταση, το οποίο καλείται να καταβάλει και αυτό 700 εκατομμύρια ευρώ. Και βλέπετε ότι καταλήγουμε κατά αυτόν τον τρόπο στα 1.500 εκατομμύρια ευρώ, τεράστιο ποσό, αλλά από το ποσό το τεράστιο αυτό μόνο τα 500 εκατομμύρια καταβάλλονται από τον οικονομικό φορέα, ενώ όλο το υπόλοιπο ποσό, περίπου 1 δισεκατομμύριο, καταβάλλεται από το κράτος και ουσιαστικά από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Ποιο είναι το μέσο κόστο, κύριε Πρόεδρε, ενό πυρηνικού ατυχήματο. Βλέπετε ότι τουλάχιστον από στατιστική πλευρά είχαμε κάποια ατυχήματα, αλλά ξέρουμε τι μα περιμένει. Είχαμε το Τσερνομπίλ και είχαμε και τη Φουκουσίμα μετά. Πέρυσι έγινε μία εκτίμηση όσον αφορά τη Φουκουσίμα, όπου ε, υπόθηκε ότι τα χρήματα που είχαν καταβληθεί ήταν 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ αν ισχύσουν οι συμφιάσεις αυτές, εμείς θα πάρουμε μόνο 1,5 ε, δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ υψηλότερα και μολονότι έχουμε πλέον και συμβάσεις δεύτερης γενιάς βάσει των στοιχείων που έχουμε η επίκριση που γίνεται αυτή, τα αρνητικά σχόλια είναι θετικά θεωρώ. επίσης από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόκληση από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Αυτό έχουν πει πάρα πολλοί αναφέροντες και αυτό ισχύει στην πράξη. Επικεντρωθήκαμε σε τέσσερα κράτη-μέλη, τα οποία είναι πολύ κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τιάνζο Βέλγιο, Γαλλία, κάτω χώρες και Γερμανία. Αν δείτε εδώ πέρα τα αριθμητικά δεδομένα, μιλάνε από μόνα τους. Η Γερμανία, από ό,τι φαίνεται, θα καταβάλει ένα ποσό των 2,5 ε, εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Γαλλία που έχει τους περισσότερους πυρηνικούς σταθμούς, 60 συγκεκριμένα, καλούνται να καταβάλουν απλώς 700 εκατομμύρια ευρώ, πολύ μικρότερο ποσό σε σχέση με τη Γερμανία. Θεωρούμε λοιπόν κύριε Πρόεδρο ότι πραγματικά Πρέπει πλέον η Ευρώπη, εσείς ουσιαστικά να πείτε ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στις διεθνείς συμβάσεις. Νομίζω πλέον ότι ισχύουν σημαντικά επιχειρήματα που κάνουν την Ευρώπη να πρέπει να αναλάβει και αυτή η δράση και μπορούμε να έχουμε ψηλότερα ποσά. Σαφώ μπορούμε. Η Ιαπωνία καταβάλει πολύ ψηλότερα ποσά. Το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε με 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ψηλό, πολύ ψηλότερο από αυτό το οποίο προβλέπεται για μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τι διεθνέ συμβάσει και ξέρετε ότι δεν έχουμε καταφέρει να προσαρμόσουμε ακόμα την νομοθεσία που υφίσταται για τις πυρηνικές καταστάσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές περιστάσεις. Αν δείτε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα τη θαλάσσια μόλυνση από το πετρέλαιο, εκεί κάθε φορά μετά από κάθε ατύχημα γίνανε και απαραίτητες νομοθετικές προσαρμογές. Για ποιο λόγο δεν έγινε κάτι τέτοιο για την πυρηνική ενέργεια. Δεν έγινε διότι εσείς ή μάλλον γίνανε προσαρμογές στο παρελθόν ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε προτάσεις στο παρελθόν και ακριβώ η ανάληψη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε και σε ανάληψη δράση σε διεθνέ επίπεδο και θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμβεί και στον τομέα τη πυρηνική ενέργεια. και νομίζουμε ότι υπάρχει πλέον η νομική βάση προκειμένου να αναλάβετε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο εσεί, τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθήσαμε να εξετάσουμε και κάποια άλλα κοινά κριτήρια όσον αφορά την εγκατάσταση, τον σχεδιασμό, την κατασκευή των πυρηνικών αυτών σταθμών. Όντω, μπορούμε εδώ πέρα να ακολουθήσουμε κάποιε βασικέ αρχέ, οι οποίε παραμένουν αρκετά ασαφεί. Και έπειτα έχουμε και τι αξιολογήσει περιβαλλοντικού αντικτύπου. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει στην πράξη ουσιαστικά εξαρτάται πάρα πολύ από τη βούληση του κάθε κράτου μέλου. Και αυτό, να θέλετε, και το γενικότερο πρόβλημα το οποίο διέπει τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν δύο οδηγίε για την πυρηνική ασφάλεια με κάποιε γενικέ αρχέ, αλλά το τι γίνεται στην πράξη εξαρτάται πάρα πολύ από την εφαρμογή που κάνουν επιτόπου τα κράτη-μέλη. Το ίδιο ισχύει και για το ζήτημα τη επιβολή τη νομοθεσία. Ακόμα και εκεί βλέπουμε ότι στα πλαίσια τη οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια προβλέπεται μια υποχρέωση υποβολή εκθέσεων από τα κράτη-μέλη, αλλά και πάλι εναπόκειται στα κράτη-μέλη να διεξάγουν ελέγχου και επιθεωρήσει. Και προβλέπονται βέβαια και τεστ αντοχή, καθώς επίσης και περιοδικέ αξιολογήσει αλλά και πάλι εγώ θα σας έλεγα να δείτε τι ισχύει για το περιβάλλον, τι ισχύει για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξουσίες επιβολής της νομοθεσίας. Για παράδειγμα, η οδηγία όσον αφορά τις εκπομπές, τις βιομηχανικές. Και εκεί πάλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες για το πώς θα πρέπει να επιβάλλεται σχετική νομοθεσία. Δυστυχώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τον πυρηνικό τομέα. Υπάρχει εδώ πέρα μια πολύ σοβαρή αναντιστοιχία. Πάλι για την πυρηνική ασφάλεια εξαρτώμεθα πάρα πολύ από τη και τις ικανότητες των κρατών μελών. Και πάλι υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν διευθετούνται, όπως για παράδειγμα τι γίνεται στην περίπτωση των μαζικών προσφυγών. Και πάλι εκεί πέρα θα έχουμε προβλήματα διεκπαιρέωσης αυτών των συλλογικών προσφυγών, αν προκύψουν. Το ίδιο ισχύει και για κάποιους άλλους τομείς. Πρέπει λοιπόν εμείς να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως θύματα. Πώς μπορούμε να λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις, να συμβάλλουμε μάλλον στη λήψη αποφάσεων ως πολίτες, ως κοινωνία των πολιτών, ως μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ξέρουμε ότι έχουμε τη σύμβαση του Άρου, τη σύμβαση του ΕΣΠΟ όσον αφορά τις, την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά θέματα και μολονότι έχει ερμηνεύσει υπέρ των θυμάτων τις δύο αυτές συμβάσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν παρόλα αυτά πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη για πυρηνικά θέματα και τελικά δεν εισακούονται. Και ξέρετε ότι υπάρχουν άδειε για συγκεκριμένη μάλλον για συγκεκριμένα πυρηνικά εργοστάσια, οι οποίε ανανεώνονται αφού ε, ολοκληρωθεί ο κύκλο ζωή του, χωρί όμω να επαναλαμβάνεται, χωρί να ανανεώνεται η μελέτη αντικτύπου. Και βέβαια αντιδρούν έντονα στο φαινόμενο αυτό πολλοί, πολλοί πολίτε. Α περάσουμε τώρα στι συστάσει. Θα μπορούσαμε να είχαμε έναν ανεξάρτητο πυρηνικό οργανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεχομένω δεν με αρέσει αυτό και θα μου πείτε ότι έχουμε την Ευρατόμ. Με Ευρατόμ, κύριε Πρόεδρε, και αυτό φαίνεται στην όλη σχετική βιβλιογραφία ότι δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει την πυρηνική βιομηχανία, να υποστηρίξει τη βιομηχανία αυτή. Να το πω κάπως ευγενικά, ο οργανισμός αυτός είναι υπέρ, πλαισιώνει, είναι με το μέρος αν θέλετε της πυρηνικής βιομηχανίας. Δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο και εσεί, οι Ευρωβουλευτέ, χρειάζεστε έναν εξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό για την πυρηνική ασφάλεια. Θεωρούμε ότι στον τομέα αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινοτική αρμοδιότητα, κύριε Πρόεδρε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο και για την κοινωνία των πολιτών. Γιατί δυστυχώ εξακολουθείτε να δίδετε πάρα πολλέ αρμοδιότητε και δικαιώματα στα κράτη-μέλη. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιες οι επιθεωρήσεις, αλλά και η δημοσίευση των εκθέσεων των επιθεωρήσεων, αν αυτές μπορούν να γίνουν, εξαρτώνται αποκλειστικά από την καλή βούληση των κρατών μελών. Νομίζουμε ότι θα μπορούσε να αναλυφθεί μια κάποια κοινοτική πρωτοβουλία για την ευθυγράμμιση των κανόνων ευθύνη, λογοδοσία και ασφάλισης, ανάληψης της ευθύνης αυτής και θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε και νομικά δεσμευτικού κανόνε όσον αφορά την επιλογή τη θέση εγκατάσταση, το σχεδιασμό και την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού. Και επίση να προβλεφθούν στην κοινοτική νομοθεσία συγκεκριμένε διατάξει σε περίπτωση συλλογικών προσφυγών. Αν γίνει κάποια τύχημα και έχουμε εκατομμύρια θύματα, εκατο... καταλαβαίνετε ότι στην περίπτωση αυτή θα έχουμε και πάρα πολλού που θα προσφεύγουν μαζικά κατά των πυρηνικών αυτών σταθμών. Όλα αυτά τα ζητήματα πιστεύω ότι θα πρέπει να διευθετηθούν, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και σας και, την, και τους συνεργάτες σας. Ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ και για το έγγραφο. Δίνω τώρα το λόγο στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο για 3-4 λεπτά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Λάβαμε την παρουσίαση μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και την σχετική μελέτη. Τι μπορώ λοιπόν να κάνω τώρα. Θα διαβιβάσουμε τη μελέτη στους αρμόδιους ε, συναδέρφους ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα τη διαβάσουν με ενδιαφέρον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο καθηγητά για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του. Να απαντήσω πολύ σύντομα. Τα καλά νέα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι πολλά από τα πράγματα που λέμε στην έκθεση είναι πράγματα που ήδη σας απασχολούν. Για παράδειγμα, ήδη εκπονείται σχέδιο οδηγίας για την εναρμόνιση των κανόνων ευθύνη. Ουσιαστικά λέμε λοιπόν, ωραία, προχωρήστε, καλά τα πάτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το θέμα της ευθύνης, θα ήθελα να προσθέσω ότι ναι, πράγματι δουλεύουμε πάνω στο θέμα αυτό. Ε, το φθινόπωρο του 2018 είχαμε σχετική μελέτη για την ευθύνη προς τρίτους ε, και θέλουμε να εξετάσουμε και την δυνατότητα ιδιωτικής χρηματοδότησης σε περίπτωση ε, κάποιου προβλήματος ε, ευθύνης στον πυρηνικό τομέα και να αυξήσουμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος. Αυτό έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις αλλά και τι μεταφορές. Και περιμένουμε μια τελική έκθεση του Συμβούλου τον Ιούλιο του 2019, Εντό του έτου δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώ έχουμε πολύ λίγο χρόνο για τη συζήτηση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια πολύ σύντομη ερώτηση Κύριε καθηγητά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες ε, οι παρατηρήσεις σας και έχετε δει όλες τις αναφορές. Συμφωνείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός ε, του Βελγίου εργάζεται με τρόπο διαφανή και ρωτώ, διότι το Σπίγκελ επανειλημμένα έχει αναφέρει ότι δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά από τον ίδιο τον οργανισμό, αλλά από άλλους φορείς. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτή την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα είμαι ειλικρινή. Είναι πολύ δύσκολο για μένα ω πανεπιστημιακό ε, να πω οτιδήποτε συγκεκριμένο γι' αυτό. Γιατί? Διότι αν δείτε πώς λειτουργεί το σύστημα, αυτή είναι ακριβώς ε, η αδυναμία του όλου συστήματος. Ε, δεν έχουμε εμεί τη δυνατότητα όπως η ΕΡΑΤΟΜ ή όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάμε κατευθείαν στο ΤΙΑΝΣ και να ελέγξουμε την πυρηνική ασφάλεια. Πρέπει λοιπόν να βασιστούμε σε ένα σύστημα εκθέσεων που υποβάλλουν οι ίδιες οι χώρες. Και μάλλον το κάνουν αυτό σωστά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει τα στοιχεία και λέει ότι το Βέλγιο πληρεί τις ε, ισχύουσες υποχρεώσεις. Άρα μπορώ να πω ότι ναι, όλα στο χαρτί είναι τέλειο. Λέω ότι το Τιάνζ είναι απόλυτα ασφαλές. Όχι, αυτό να μην το παραθέσετε ως δικά μου λόγια. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Έτσι λειτουργεί το σύστημα και Γι' αυτό διστάζω να κάνω πολύ σαφείς δηλώσεις πάνω στο θέμα αυτό. Ελπίζω να καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Και περνάμε τώρα σε συγκεκριμένες αναφορές. Δόκτωρ Τιμ Γκρίτεμαγερ και Κρίστελ Σλέμπους από τη Γερμανία. Δύο αναφορές σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Τιόνς 2. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Τέσσερα λεπτά ο καθένας. Γκίτε Μάιρ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Αναφορών, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλώ στο όνομα της ε, της ε, συλλογικής ε, δράσης ε, που περιλαμβάνει 100 χώρες και περιφέρειες από το Λουξεμβούργο, τις 100 χώρες και τη Γερμανία. Έχουμε ανησυχίες ως πολίτες της Ένωσης. Αμφιβάλλουμε όσον αφορά την εκτίμηση της Βελγικής Αρχής Πυρηνικής Ενέργειας σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Τιόνς 2. Ο νέος Υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου δεν ε, βλέπει ως ρεαλιστική λύση την εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας μέχρι το 2025. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν στρεφόμαστε κατά ε, κάποιου κράτους μέλους. Αντιθέτως, σεβόμαστε απόλυτα την, ε, το κυρίαρχο βασίλειο του Βελγίου. Ωστόσο, έχουμε την πυρηνική ένωση, την πυρηνική κοινότητα, και στο προήμιο αυτής ε, αναφέρεται ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια για να αποκλειστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι για τον πληθυσμό. Υπάρχουν όμως ρογμές στον πυρηνικό αντιδραστήρα TIONS-2, κάτι που οδηγεί σε αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα μόνο. Υπάρχουν πολλές ρογμές, των οποίων ε, την αιτία δεν γνωρίζουμε. Έχουν, έχει αυξηθεί ο αριθμός αυτών και οι ρογμές που ήδη έχουν διαπιστωθεί έχουν ε, μεγαλώσει. Ε, υπάρχουν ε, επιτροπές εμπειρογνωμόνων που δεν δηλώνουν σαφώς ότι είναι ασφαλής ο αντιδραστήρας. Για παράδειγμα, το, 2000, το Ιανουάριο του 2013 διαπιστώθηκε διαρροή υδάτων στο μη πυρηνικό τμήμα του αντιδραστήρα. Ο φορέας ε, λειτουργίας διαπίστωσε επίσης ότι ε, είχε αυξηθεί η θερμοκρασία των ε, υδάτων ψήξης. Το καλοκαίρι του 2016 υπήρχαν προβλήματα με μια αντλία στο πυρηνικό τμήμα και διακόπη η λειτουργία του αντιδραστήρα το φθινόπωρο του 2018 αποφασίστηκε να κλείσει ο αντιδραστήρας. Ε, διαπιστώθηκε ένα πρόβλημα σε ένα διπλανό κτίριο και αυτό μάλιστα θεωρήθηκε περιστατικό ε, κλάσης 1. Θεωρήθηκε όμως ότι μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία το 2019 το αντιδραστήριο. Τον Οκτώβριο του 2018 το Der Spiegel ανέφερε πολλά, πολλά μικρά περιστατικά ε, τα οποία δεν είχε αναφέρει ο φορέας λειτουργίας ε, του αντιδραστήρα και μάλιστα 11 ε, ανθρώπους ε, που είχαν εκτεθεί σε ραδιενέργεια. Έχουμε την αρχή της προφύλαξης που είναι βασική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου. Ε, δεν ε, μπορούν ε, να αποδεχτούν οι πολίτες μια τέτοια στάση. Η Κομισιόν λέει ότι η υποβολή των εκθέσεων από πλευράς του Βελγίου ήταν ικανοποιητική, αλλά αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Λείπουν κάποια πολύ σημαντικά έγγραφα. Συγκεκριμένα δεν υπάρχουν τα εξή στοιχεία. Έκθεση της Εθνικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, του 2012 η γραπτή αιτιολόγηση της επαναλειτουργίας του σταθμού ε, του 28 Ιανουαρίου του 2016 ε, έκθεση της Μπελφάου του 2015 καθώς και ε, συζητήσεις το 2015 ανάμεσα στην ΦΑΝΚ και την Ελεκτραμπέλ. αναφέρεται ότι είναι διαφανείς ε, οι οργανισμοί αυτοί, αλλά πώς είναι αυτό δυνατό τη στιγμή που υπήρχαν 250 περιστατικά τα οποία ε, είχαν συγκαλυφθεί. Η διασφάλιση της ε, ποιότητας μπορεί να διασφαλιστεί μόνο αν υπάρχει απαραίτητη τεκμηρίωση από πλευράς του Βελγίου. Ζητάμε από την Επιτροπή Αναφορών να μην κλείσει την αναφορά αυτή ε, την παρακαλούμε επίσης να στείλει επιστολή στη, στο Βέλγιο καθώς και στον ε, φορέα εποπτείας ΦΑΝΚ του Βελγίου. Θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική τεκμηρίωση σχετικά με την ασφάλεια του πυρηνικού αντιδραστήρα. Η Κομισιόν καλό θα ήταν να καλέσει ε, το Βέλγιο να υποβάλει τα έγγραφα που λείπουν στην τεκμηρίωση σχετικά με την ασφάλεια του σταθμού Τιόνς 2. Βλέπουμε παραβίαση της ε, αρχής της προφύλαξης ε, που θεσπίζεται στην συνθήκη Euratom. Πιστεύουμε ότι πρέπει κάτι να γίνει στην περίπτωση αυτή και δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρηθεί ε, ότι έχει κλείσει η αναφορά αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέσσερα λεπτά η κυρία Κρίστελ Σλέιμπους. Έχω υποβάλει αυτή την αναφορά ώστε να μην, να μπορεί το κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει αν θα πρέπει να κλείσει ένας πυρηνικό σταθμός ή όχι. Υπάρχει ευρωπαϊκή εποπτεία, αλλά η απόφαση για κλείσιμο ε, πυρηνικού αντιδραστήρα εναπόκειται στο κάθε κράτος μέλος ε, και μάλιστα συχνά στον ε, φορέα λειτουργίας του σταθμού. Η Επιτροπή του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον, πάντα λέει ότι όλα είναι σωστά τεκμηριωμένα και ότι εξετάζεται προσεκτικά το τι γίνεται. Μάλιστα, είπε κατά λέξη ότι οι υπηρεσίες της Κομισιόν ε, εξετάζουν τις στοιχείες πυρηνικής ενέργειας ε, όσον αφορά τους πυρηνικούς σταθμούς ε, στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του σταθμού Τιόνς 2. Αυτό όμως δεν ισχύει. Δεν αποκλείεται τα οικονομικά συμφέροντα του κάθε κράτους μέλους να θέτει σε κίνδυνο την προστασία του πληθυσμού. Όσον αφορά τον σταθμό Τιόν 2, επανειλημμένα έχουμε δει ότι αποσιωπήθηκαν ε, κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, είχαμε 11 ανθρώπους που εκτέθηκαν στην ραδιενέργεια και Πράγματα τα οποία δεν έχουν όπως ακριβώς παρουσιάζονται. Το γερμανικό περιοδικό Spiegel τον Οκτώβριο του 2018 ανέφερε 250 νέα περιστατικά όσον αφορά τον σταθμό Tions 2. Ο φορέα ΦΑΝΚ δεν φαίνεται να είναι ανεξάρτητος. Δίδεται μάλλον η εντύπωση ότι προσπαθεί να κρύψει πράγματα. Ε, χάπια ιωδίου, όπως ε, ήδη έχει γίνει, που μοιράζονται στον πληθυσμό ε, ως πρόληψη σε περίπτωση ενός ατυχήματος, δεν είναι μόνο κάτι γελίο, δείχνει ε, την ε, αμηχανία των αρχών. Δεν Όπως επίσης δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ε, τα, στοιχεία, ε, τα, τα σχέδια επίγουσα ανάγκη. Ε, σκεφτείτε εκένωση μια πόλη σαν το Άχεν. Στο, στην Τιάνς βλέπουμε όλο και νέες ρογμές και είναι δυνατόν να παρατείνουμε συνέχεια τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού σαν να είναι απλά ένα παλιό πλυντήριο που έχει χαλάσει. Δεν θέλουμε πια να βασιζόμαστε στην όλο και λιγότερο πιθανή τύχη μας ε, να μην συμβεί κάτι τρομερό. Η Γερμανία μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα αποφάσισε να εγκαταλείψει την ε, πυρηνική ενέργεια, ενώ ε, από τους Ιάπωνες περιμένουν ακόμα να συνεχίσουν να ζουν σε ένα έδαφος με πολύ υψηλή σεισμικότητα, όπου υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί. Δεν αναφέρεται η πρόληψη με χάπια ιωδίου. Βλέπουμε όλο και περισσότερες ρογμές. Ε, ακούμε ότι όλα είναι πάρα πολύ διαφανή, παρότι περιστατικά ε, δεν σχολιάζουν μέχρι να διαρρεύσουν ε, στο κοινό. Ενώ οι γραπτές ερωτήσεις παραμένουν αναπάντητες. Η Κομισιόν συνεχίζει να βασίζεται στα στοιχεία της ΦΑΝΚ, παρότι εμπειρογνώμονες έχουν φτάσει σε ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ότι δυστυχώς και σίγουρα όχι αμέσως δεν μπορούμε να ζητήσουμε το κλείσιμο όλων των πυρηνικών σταθμών στην Ευρώπη. Δεν έχει γίνει ο απαραίτητο προγραμματισμός για κάτι τέτοιο. Και δυστυχώς η Αυστρία που ποτέ δεν είχε πυρηνικού σταθμούς αποτελεί εξαίρεση. Αυτό που ζητάμε όμως ε, είναι κλείσιμο των παλιών σταθμών ε, όπως είναι ο Τιόνς 2, με μία όσο γίνεται ανεξάρτητη ευρωπαϊκή εποπτεία. Σας ευχαριστώ. Uh, Και εγώ σας ευχαριστώ. Δίνω πάλι το λόγο στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Ανέτα Σέιτσκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που έκαναν τον κόπο να έρθουν εδώ και να παρουσιάσουν την κατάσταση και τις ανησυχίες τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να τονίσει ότι ακούει ε, και παρακολουθεί τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών και ιδιαίτερα όσον αφορά ε, την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού Τιόνς. Όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια, θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η απόφαση για την μακροπρόθεσμη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και η πυρηνική ασφάλεια βρίσκεται στα χέρια ε, των φορέων λειτουργίας ε, των πυρηνικών σταθμών που εποπτεύονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ωστόσο, η πυρηνική ασφάλεια και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στόχος μας είναι να φροντίσουμε να παράγεται πυρηνική ενέργεια με σεβασμό του πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια. Γι' αυτό οι υπηρεσίες ε, της Επιτροπής παρακολουθούν ε, την ε, συμμόρφωση του Βελγίου με την σχετική νομοθεσία συμπεριλαμβανομένη στις λογοδοσίες του Φορέα Λειτουργίας και της διασφάλισης από πλευράς του της ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά θέματα πυρηνικής ασφάλειας, όπως και τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και ιδιαίτερα του TIONS 2. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με κάποια στοιχεία, σχετικά με την πρώτη έκθεση ομοτήμων την πρώτη αξιολόγηση ομοτήμων που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αναθεωρημένη οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια. Ο στόχος, ε, ε, το, το κύριο θέμα εδώ πέρα ήταν η ασφάλεια και η ηλικία των πυρηνικών σταθμών. Το Βέλγιο συμμετείχε πλήρως ε, στην όλη προσπάθεια. Ως τμήμα της προσπάθειας να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών πάνω στο θέμα αυτό, οργανώθηκε μια δημόσια εκδήλωση για το θέμα αυτό πέρσι στις 3 Μαΐου. Από 14 ε, ε, έως 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ε, μια, ένα σεμινάριο αμοιβαίας αξιολόγησης, αξιολόγησης ομοτήμων, ενώ παρουσιάστηκαν τα τελικά στοιχεία στην ιστοσελίδα τον Οκτώβριο του 2018 και παρουσιάστηκαν επίσης σε μια δημόσια εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Η Άνσακ ε, ετοιμάζει ε, μια επισκόπηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και με βάση αυτόν τον πίνακα όλες οι χώρες που συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένου και του Βελγίου, ετοιμάζουν τα δικά τους εθνικά σχέδια δράσης. Στόχος είναι να εφαρμοστούν ε, τα συμπεράσματα αναχώρα μέσω των σχεδίων αυτών. Αναμένεται ε, να παραληφθούν Σεπτέμβριο του φετινού έτους τα σχέδια αυτά. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει επίσης να σας ενημερώσει ότι το θέμα το, της ε, μεγάλης ηλικία των πυρηνικών εργοστασίων στην Ευρώπη θα συζητηθεί και σε ένα άλλο βήμα. Στην ε, στο επόμενο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί φέτος τον Απρίλιο στην Πράγα. Είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερομένους η εκδήλωση αυτή ε, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, ε, θεσμικών οργάνων, ε, ρυθμιστών ενέργειας και της κοινωνίας των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Τώρα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν το λόγο. Κύριε Σκόχ, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ω Ευρωβουλευτή ε, του Άχεν, με ρωτάνε συχνά γιατί η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα για το ΤΙΑΟΣ Και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία αυτή και τι σχετικέ αναφορέ που έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε εδώ σήμερα, καθώ και για τη μελέτη που μπορέσαμε να δούμε, διότι μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να συζητήσουμε εδώ το θέμα αυτό οι κανόνες, οι συνθήκες και διεθνείς συμβάσεις που ίσχυαν μέχρι τώρα δεν, αρκούν. Χρειαζόμαστε ένα ε, αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για πυρηνικά εργοστάσια όπως είναι το TIANS που ε, προκαλεί ανησυχίε σε πολλού ανθρώπους ε, τη περιοχής, της ευρύτερης περιφέρειας, ακόμα και τη δική μου οικογένεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν ασφάλεια και χρειαζόμαστε αποτελεσματικούς ελέγχους και όχι μόνο ελέγχους που να φαίνονται αποτελεσματικοί στο χαρτί, αλλά που στην πραγματικότητα δεν είναι. Το Τιόνζ είναι καλό παράδειγμα που δείχνει ότι Χρειάζεται να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται να κοιτάξουμε πέρα από τα προσωπικά και εθνικά μας συμφέροντα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε όλους τους ανθρώπους ε, στην περιοχή ε, του Ρήνου και ε, και σε άλλες περιοχές άλλωστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ε, κύριε κυρία Σλέπους. Έχουμε το εξής μήνυμα για σας. Στηρίζουμε τις αναφορές σας. Ε, προτείνω να παραμείνουν ανοιχτές οι αναφορές αυτές, ε, όπως προτείνατε, και προτείνω επίσης να σταλεί ε, επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος είπε ότι θα είναι χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των παλαιών ε, πυρηνικών σταθμών, ιδιαίτερα στο Βέλγιο και ιδιαίτερα για τον σταθμό Τιόνς 2. Θα στείλουμε επιστολή στο, στη βελγική κυβέρνηση με το ίδιο αίτημα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, και στο Βέλγιο, διότι δεν είναι πολύ σαφής ε, ο ρόλος ε, του Οργανισμού ε, Πυρηνικού Ελέγχου. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να στείλουμε επιστολή στις βελγικές αρχές για το θέμα αυτό, γιατί δεν είναι πολύ σαφής η κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ναι, φυσικά θα κάνουμε αυτό που προτείνατε. Δίνω το λόγο για δύο λεπτά στον κύριο Γκρίτεμαγερ και την κυρία Σλέβους. Δύο λεπτά, αν θέλετε το λόγο. Ναι. Ελπίζω, εάν συζητηθεί η συνθήκη Euratom τον Μάρτιο με αφορμή το Brexit, να γίνουν και οι απαραίτητες τροποποιήσεις όσον αφορά ε, τους ε, πυρηνικούς σταθμούς. Θεωρώ πολύ σημαντικό όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί ηλικία 40 ετών που ακόμη λειτουργούν και με τους οποίους συναντάμε πολλά προβλήματα να έχουν καλύτερη εποπτεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ναι, παρακαλώ, κύριε Κρούτεμαγερ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο. Ε, Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σα. Ε, σα ευχαριστούμε που αφήνετε ανοιχτή την αναφορά αυτή και για τι περαιτέρω εργασίε. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε δύο άλλε αναφορέ από την Ισπανία. Αναφορά 434 σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό στην πόλη Μπούργος και την αναφορά 0312 για το ίδιο θέμα. Από ό,τι με ενημερώνουν είναι παρόν ο αναφέρον. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 25 Απριλίου του 2017 σε αυτή την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μίλησα για, την, ε, το οριστικό κλείσιμο του πυρηνικού εργοστασίου της Γκαρόνια. Αλλά η Ισπανική κυβέρνηση μίλησε για μια νέα παράταση της λειτουργίας του. Ε, μιλάμε για ένα πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο είχε κλείσει από το 2012 και όλες οι επιχειρήσεις που το εκμεταλλεύονταν αυτό το εργοστάσιο ε, δεν είχαν κάνει τις ε, εγγύησεις, τις ε, απαραίτητες επενδύσεις, για την ασφάλεια ε, δεν είχαν ενημερώσει το κοινό κτλ. Ε, δεν ενημέρωσαν κανένα και ούτε σε ενδιαφέρει να το κάνουν. Η αναφορά έμεινε ανοιχτή και ζητήσαμε την κυβέρνηση της Ισπανίας να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η απόφαση δύο μήνες ε, μετά από την Ισπανική κυβέρνηση ήταν να κλείσει οριστικά το πυρηνικό εργοστάσιο της Σάντα Μαρία Ντεκαρόνια και παρόλα αυτά σε καμία περίπτωση το δίκτυο ηλεκτροδότης τη Ισπανίας δεν επηρεάστηκε. Ε, θεωρήθηκε ότι ξεκίνησε η περίοδος διάλυσης και η αποκατάσταση της ε, ζώνης αυτής, ε, της κοιλάδας στον Παλίνα. Αλλά ξεκίνησε μια περίοδος τότε αβεβαιότητας, παραπληροφόρησης, έλλειψης διαφάνειας, αλλαγής κυβέρνησης, καθυστερήσεων σε αποφάσεις κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά τα θέματα της συνθήκης Euratom, όπου οι φορείς και οι οι εταιρείε καθώς και η Ισπανική κυβέρνηση δεν τηρούν. Ε, σε καμία περίπτωση δεν λήφθη υπόψη ότι το όργανο που υποτίθεται θα ήταν ανεξάρτητο για την αξιολόγηση της πυρηνική κατάστασης στην Ισπανία, ε, το οποίο είναι το CSN, ε, το οποίο είναι ένα όργανο που έχει πολιτική απόχρωση και δεν έχει δώσει ε, σωστές ε, πληροφορίες. Τίθονται λοιπόν τα επόμενα ερωτήματα. Έχουμε την οδηγία 2011-70 για τη διαχείριση με ασφαλή τρόπο των ραδιενεργών καταλήπων, που είναι πολύ σαφή. Μιλάει για τον τρόπο που λαμβάνονται οι άδειε για να λειτουργήσει μια επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει τη συνθήκη Euratom. Ε, και οι εταιρείε οι οποίε χειρίζονται ραδιενεργά πόλητα θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν, να εκμεταλλευτούν και να διαλύσουν με ασφαλή τρόπο ε, μια πυρηνική εγκατάσταση. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι καμία από τις εταιρείε που λειτουργούν στην Ισπανία στον πυρηνικό τομέα δεν μπορούν να αποδείξουν, καμία λέω, ε, άρα δεν σέβονται την ε, συνθήκη της Euratom, ε, ότι σέβονται τους κανόνες ε, στα πυρηνικά εργοστάσια, ούτε καν στο, στο Σάντα Μαρία Γκαρόνια. Στην Ισπανία λοιπόν οι εταιρείε εκμεταλλεύονται, αλλά δεν αποκαθιστούν. Ε, και ποιο αποκαθιστά η Ενρέσα, που είναι μια δημόσια εταιρεία η οποία κάνει τη βρώμικη δουλειά και στην περίπτωση τη Γκαρόνια ε, μιλάμε για 480 εκατομμύρια ευρώ τα οποία ε, εκταμιεύτηκαν από το Γενικό Κρατικό Προπολογισμό για να καθαρίσει η Γκαρόνια, ε, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τη διαχείριση των καταλήπων. Η Ισπανία είναι μία από τι ευρωπαϊκέ χώρε με το υψηλότερο κόστο ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι με βάση την έκθεση που έγινε η οργάνωση ε, για τι ε, περιβαλλοντικέ επιστήμε για την ενεργειακή φτώχεια, ε, αποδείχθηκε το 2018 προκύπτει ότι 19 εκατομμύρια άτομα, το 41% του πληθυσμού της Ισπανίας, ε, πάσχει από την ε, λεγόμενη ενεργειακή φτώχεια, πολύ παραπάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι φορείς εκμετάλλευσης της πυρηνικής ενέργειας στην Ισπανία, ε, μιλάμε για 10 εταιρείε που μολύνουν τη χώρα μας, στην πραγματικότητα απλώς κερδοσκοπούν από το πυρηνικό εμπόριο και το κράτος ε, απλώς κάνει τη βρώμικη δουλειά, καθαρίζει ας πούμε ε, τις βρωμιές τους. Ε, η Ευρωπαϊκή Συνθήκη Euratom για την Ευρωπαϊκή Ενέργεια στο άρθρο 21 λέει ξεκάθαρα ότι τα ραδιενεργά απόβλητα καθώς και το, ε, τα χρησιμοποιημένα ε, πυρηνικά καύσιμα πρέπει να περιοριστούν και να απομακρυνθούν από την επαφή με τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Ε, χρειάζονται μέτρα για να προστατεύσουμε από τους κινδύνους και, τις, ε, ε, τη ραδιενέργεια, για να προστατεύσουμε λοιπόν τους ανθρώπους και την υγεία καθώς και το περιβάλλον. Χρειάζονται μέτρα που προβλέπουν την οριστική αποθεματοποίηση σε, από, σε ειδικές εγκαταστάσεις και την προσωρινή αποθεματοποίηση ε, για ένα συγκεκριμένο ε, χρόνο ε, ως μια προσωρινή λύση μέχρι να βρεθεί η οριστική λύση. Στην Ισπανία καμία κυβέρνηση δεν μπόρεσε να ε, ρυθμίσει το θέμα της αποθεματοποίησης. Στην περίπτωση της Γκαρόνια, στην πραγματικότητα αυτά τα κατάλοιπα τα αφήνουμε ελεύθερα, εκτεθειμένα στο κλίμα, στον αέρα, ε, και μάλιστα είναι, βρίσκονται κοντά στον ποταμό Εύρο ε, για ε, επαόριστο. πρέπει να, να προσθέσουμε ότι έγινε ένα project, το μοναδικό project για την οικοδόμηση μιας κεντρικής αποθήκης στην Ισπανία με την ιδέα όμως ότι θα κλείσουν όλα τα πυρηνικά εργοστάσια της Ισπανίας όσα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους της 4 ετίας ε, χωρίς να γίνει ε, όμως καμία τροποποίηση ή επέκταση της ε, διάρκειας ζωής τους. Άρα, τι μπορούμε να πούμε, ότι δεν σεβόμαστε την ε, οδηγία 2009-71 σε ό,τι αφορά το, ε, τις διατάξεις 12 για την ε, υποχρέωση προσωρινής και οριστικής αποθεματοποίησης. Ε, την οδηγία 2011-70 στα στις διατάξεις 19, 20, 21, 30, 31 και τα άρθρα 5, 7, 10 και 11 σε ό,τι αφορά το σχέδιο, τις προθεσμίες, τη διαφάνεια, το κόστος και την χορήγηση των αδειών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτιάξουμε ένα σχέδιο ανάκτησης της μολυσμένης ζώνης γιατί συνεισφέρει στο ενεργειακό σύστημα της Ισπανίας. Ε, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ε, με καθαρές ενέργειες, ε, Θέλουμε ε, βιώσιμη ανάπτυξη για την περιοχή, δηλαδή για την επαρχία Μερινδάδες και όχι την ε, δαμόκλειο σπάθα της υδρορογμάτευσης, ε, τα ορυχεία, της ε, τα λατομεία, ε, τα οποία λειτουργούν γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο τη Σαντα Μαρία Δεκαρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απαιτήσει άμεσα ε, την, ε, το να σεβαστεί η κυβέρνηση της Ισπανίας ε, την συνθήκη της Euratom. θα πρέπει να προστατεύσουμε τα άτομα, θα πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Κύριε Σιέκα, έχετε πάλι το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Αναφέροντα. Λοιπόν, Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η επιλογή που γίνεται για τους ενεργειακούς πόρους και για το αν θα πρέπει να λειτουργήσει ή όχι πυρηνικός σταθμός εναπόκειται καταρχάς σε κάθε κράτος μέλος. Από τις γενικές πληροφορίες που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι η λειτουργία του σταθμού Σάντα Μαρία Ντεγκαρόνια δεν πρόκειται να επεκταθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει πληροφορίες σχετικά με περαιτέρω επενδύσεις επαντηλειτουργίας του σταθμού αυτού. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αν το κράτος μέλος αποφασίσει να επεκτείνει τη λειτουργία του πυρηνικού αυτού σταθμού ή οποιοδήποτε άλλο πυρηνικού σταθμού, θα πρέπει να πληρεί τα κριτήρια πυρηνικής ασφάλειας όπως προβλέπονται από τη συνθήκη και τη δευτερογενή νομοθεσία. Το παράγωγο δίκαιο μάλλον. Όσον αφορά τώρα τον διαχειρισμό του παροπλισμού ενός πυρηνικού σταθμού, κάθε κράτος μέλος οφείλει να έχει ένα εθνικό νομοθετικό όσον αφορά τα ρεδινεργά απόβλητα και τα χρησιμοποιημένα, ξαντλημένα απόβλητα. Αυτό προβλέπεται από την συνθήκη Ευρατόμου. Επίσης, όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια, τη βασική ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια ενός, μιας πυρηνικής εγκατάστασης φέρει ο κάτοχος της άδειας, δηλαδή ο φορέας εκμετάλλευση στο πλαίσιο της λειτουργίας της ρυθμιστικής αρχής. Αυτό προβλέπεται και στην κοινοτική οδηγία 71-2009 όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων. πάνω η Ισπανία, όπως οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος οφείλει να μεταφέρει καταλήλω στην δική της νομοθεσία τις δύο αυτές κοινοτικέ οδηγίες και να εφαρμόσει τις απα... απαιτήσει των οδηγιών αυτών και θα πρέπει βέβαια να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ μεταφέρθηκαν και πώ εφαρμόζονται οι δύο αυτέ οδηγίε. Επίση, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στα πλαίσια της συνθήκης Ευρατών τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιτηρούν το επίπεδο της ραδιενέργειας στον αέρα, το έδαφος, το νερό, καθώς επίσης και στα τρόφιμα. Και πάλι θα πρέπει να ενημερώνουν καταλήλως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να έχουν τα απαραίτητα μέσα προκειμένου αποτελεσματικά να μπορούν να κάνουν αυτές τις μετρήσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κι εμείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Μαρτσερέζη πρώτος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ε, αναφέροντα για την ε, παρέμβασή του. Χαίρομαι καταρχάς που έκλεισε αυτό το εργοστάσιο της Γκαρόνια ε, από την τελευταία αναφορά που έγινε μέχρι σήμερα. Αυτό είναι καλό νέο, γιατί ήταν εργοστάσιο το οποίο ήταν πολύ δαπανηρό, ήταν περιττό και πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση, που είναι η φάση, μια φάση περίπλοκη για, την, για τον παροπλισμό της εγκατάστασης αυτής. Έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα που σχολίασε ο αναφέροντας και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς, είναι η έλλειψη πληροφορίας, δεν είναι καινούριο, το είδαμε και προηγουμένως με τη μελέτη που μας παρουσιάστηκε. Υπάρχει ένα πρόβλημα ανεξαρτησίας ε, των ατόμων που δίνουν πληροφορίες ε, για θέματα πυρηνικής ενέργειας. Έχουμε δημάρχους σε αυτήν την περίπτωση, έχουμε τους πολίτες, έχουμε κοινωνικούς παράγοντες που δεν είναι ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει για το πυρηνικό αυτό εργοστάσιο. Ε, είναι μια μεγάλη μαύρη τρύπα, δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικές η ανεπάρκειες όσον αφορά τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Από ό,τι φαίνεται η Ισπανία δεν καλύπτει τις διατάξεις και τα όσα απορρέουν από τις δύο κοινοτικέ οδηγίες. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν καν κεντρικές μονάδες διαχείρισης και επεξεργασίας των πυρηνικών αποβλήτων. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει οι αναφορές αυτές να παραμείνουν ανοιχτές, να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες μέσω επιστολής από τις αρμόδιες αρχές να μας δώσει περισσότερα στοιχεία επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν έχει λάβει δηλαδή ενημέρωση και αυτή από τις Ισπανικές Αρχές και θεωρώ ότι ε, θα πρέπει πλέον όλη αυτή η περιοχή πάνω από τον Μπουργκος να αρχίσει να επενδύει περισσότερο σε βιώσιμες μορφές ενέργειας. Ας εγκαταλείψουμε πλέον αυτές τις μη βιώσιμες μορφές ενέργειας. Ας εγκαταλείψουμε την υδρορογμάτωση, ας εγκαταλείψουμε τα λατομία και επιτέλους ας προωθήσουμε καθαρές μορφές ενέργειας. Ας αποστείλουμε λοιπόν μία επιστολή στις αρμόδιες αρχές για όλες τις παραβιάσεις που έχουμε δει στην περιοχή της Γκαρούνια. Η κυρία Ελμπιόλ Γκουθμάν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάθε φορά που εστιαζόμαστε στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας στην Ισπανία, αυτό το οποίο συνειδητοποιούμε είναι ότι υπάρχουν πολλές παρατυπίες, έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη πληροφοριών και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και σε αυτή την αναφορά και θα φανεί και στις μελλοντικές, σας το υπόσχομαι. Στην αναφορά για παράδειγμα για το παλωμάρες που θα ακούσουμε σε λίγο, αλλά και λίγο αργότερο θα συζητήσουμε το ζήτημα του El Καμπρίλ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο ανακύπτει συνεχώς όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια στην Ισπανία. Έλλειψη πληροφοριών, αυτοσχεδιασμοί, ημίμετρα. Και όλα αυτά οφείλονται στο ότι έχουμε όλες αυτές τις μεταπηδήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων προς ιδιωτικές εταιρείες. 16 το αριθμό από το Λαϊκό Κόμμα καθώς επίσης και από το Σοσιαλιστικό Κόμμα οι οποίοι έχουν περάσει στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων ενεργειακών εταιριών. Εν λοιπόν τι βλέπουμε. ουσιαστικά βλέπουμε ότι το οικονομικό κέρδος θεωρείται πολύ πιο σημαντικό από το συλλογικό συμφέρον. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, ιδιαίτερα σημαντικό για την ανθρώπινη υγεία, αλλά και γενικότερα για την υγεία του πλανήτη μας. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της συνθήκης Ευρατόμ. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και θα ζητούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς ε, τη διαδικασία παροπλισμού του Γκαρούνια και να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται με τα πυρηνικά απόβλητα και να μας ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε παρατυπία. Συντοποιούμε ότι όλα αυτά αποτελούν εθνική αρμοδιότητα της Ισπανίας, ο παροπλισμός κυρίως δηλαδή, αλλά νομίζω ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει την ευθύνη της ενημέρωσης και φέρει επίση την ευθύνη της παρακολούθησης της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας και της συνθήκης Ευρατόμ. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτηρήσει ιδιαίτερα επισταμένος την όλη διαδικασία. Έγινε μια ερευνητική, διερευνητική ε, αποστολή στην Ισπανία σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια και τα πυρηνικά κατάλοιπα. Έχουμε αυτή την ε, αναφορά, έχουμε άλλες δύο σχετικές αναφορές με άλλα ζητήματα, συναφή Υπάρχουν πάρα πολλέ λοιπόν σχετικέ αναφορέ που έχουν να κάνουν με τον ενεργειακό τομέα και την πυρηνική ενέργεια στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Κυρία Βαλίνα. Δεν θέλετε να μιλήσετε. Κύριος Μπενίτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήξερα να πάρω το λόγο να μην το πάρω, γιατί δεν γνωρίζω την αναφορά. Ε, δεν ξέρω, άκουσα απλώ τι είπε, αλλά τέλο πάντων αναφέροντα, ε, μου τα εξήγησε πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Γιατί παίρνω το λόγο, λοιπόν. Μετά την απάντηση τη Κομισιόν, αισθάνομαι αναγκασμένο να πάρω το λόγο. Θα ήθελα περισσότερε πληροφορίε. Ξέρουμε ότι το πυρηνικό εγκροστάσιο τη Γκαρόνια σταμάτησε να λειτουργεί το 2012. Έκτοτε, η... ακούσαμε διάφορες απειλές ε, για επανέναρξη της λειτουργίας ε, του ε, εργοστασίου αυτού, ε, αλλά σταμάτησε, σταμάτησε οριστικά, αποφασίστηκε να μην λειτουργήσει ενώπιον της πίεσης από τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει το 2019 και δεν έχει γίνει σοβαρός παροπλισμός του, της εγκατάστασης αυτής. Αυτό που μου φαίνεται πολύ σοβαρό για αυτή την κατάσταση είναι ότι ο παροπλισμός που προβλέπεται δεν γίνεται με σεβασμό τη συνθήκη Euratom, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η, εταιρεία η οποία ήταν αρμόδια και εκμεταλλεύτηκε τον σταθμό αυτό, δεν ασχολείται με τον παροπλισμό του, της εγκατάστασης, ασχολείται μια δημόσια επιχείρηση. Βλέπουμε ότι τα κέρδη είναι ιδιωτικά, ενώ το κόστος του παροπλισμού είναι δημόσιο. Βαραίνει το δημόσιο κορβανά. Αυτό είναι τελείω άδικο. Πολύ σοβαρό και πολύ άδικο. Διερωτώ με λοιπόν, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα, δεν θέλει να παίξει το ρόλο της ως θεματοφύλακα των συνθήκων. Ακόμα ένα ερώτημα και θα τελειώσω. Νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί προγράμματα μετάβαση και μάλιστα δίκαιη μετάβαση. Έχουμε εδώ πέρα μία μετάβαση. Μιλάμε για μία περιοχή όπου υπήρχε ένα ε, πυρηνικό εργοστάσιο που λειτουργούσε, το οποίο σταμάτησε και έπρεπε να παροπληστεί. Και μιλάμε για μία ε, μετάβαση η οποία πρέπει να γίνεται δίκαιη. Δηλαδή η επιχείρηση είναι αυτή που πρέπει να πληρώσει για τον παροπλισμό. Θα ήθελα λοιπόν να μου δοθούν περισσότερα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν πρέπει, δεν πρέπει να προσφύγετε εναντίον των Ισπανικών αρχών. Εν πάση περιπτώσει, αν όχι να προσφύγετε εναντίον του, τουλάχιστον να πάρετε περισσότερε πληροφορίε από την Ισπανία. Αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο, ο πυρηνικό σταθμό, δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 70 και έκλεισε το 2012. Το 2006 είχαμε κάποιε αμφιβολίε, γι' αυτό σκεφτόμασταν μήπω θα πρέπει να τον ξανανοίξουμε αυτό το σταθμό ή όχι. Τελικά αποφασίστηκε να κλείσει. Τα σχέδια όμως τα τηρούμε, γιατί ο παροπλισμός ε, θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμεινο του 2019 και είναι μια δύσκολη διαδικασία που παίρνει πάνω από 10 χρόνια. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι λέτε ακριβώς. Η Κομισιόν εποπτεύει την υλοποίηση αυτών των σχεδίων και το σεβασμό των ευρωπαϊκών οδηγιών. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην Κομισιόν. Εγώ δεν καταλαβαίνω, εφόσον σεβόμαστε τα σχέδια ε, εφόσον υπάρχει νομιμότητα, εγώ θα έλεγα να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Εάν κάτι δεν γίνεται καλά, να έρθουμε εδώ πέρα και να παραπονεθούμε. Αλλά να παραπονεθούμε προληπτικά, α πούμε, μπα και γίνει κάτι στραβό, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Η Κομισιόν είπε ότι όλα γίνονται όπω πρέπει, με βάση τον νόμο. Είμαστε εμπρόθεσμοι, επομένω δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Δεν αθετεί το Ισπανικό κράτο τι υποσχέσει του. Επομένω, κατά την άποψή μου, πρέπει να κλείσει αυτή η αναφορά. So I think can make resume in, in, in three points. Λοιπόν, να συνοψίσουμε σε τρία σημεία. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, είναι αναγκαίο και είναι και δυνατό να αποστείλουμε μία επιστολή προς τις Ισπανικές Αρχές και να τους ζητήσουμε για περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνούμε με αυτό. Πολύ ωραία. Δεύτερον, Νομίζω ότι είναι θεμητό να αποταθούμε εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσουμε και από την Επιτροπή περισσότερες πληροφορίες. Και στη συνέχεια μπορούμε να ταθούμε υπέρ της μίας της άλλης σύστασης, να μην ανοιχτεί η αναφορά ή να την κλείσουμε. Να ψηφίσουμε, τι λέτε. Ποιο είναι υπέρ του να μείνει ανοιχτή αναφορά μετά τα δύο αυτά βήματα τα οποία περιέγραψα. Ποιο είναι υπέρ του να μείνει ανοιχτή αναφορά. Τρει. Ποιο θέλει να κλείσει αναφορά. Δύο. Λυπάμαι, αλλά στην περίπτωση αυτή η ψήφος του Προέδρου είναι καθοριστική. Είμαι υπέρ του να κλείσει αναφορά εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι κρίμα, κρίμα που κλείνει η αναφορά αυτή. Πραγματικό κρίμα. Νομίζω ότι παραπληροφορούμε και την Επιτροπή των Αναφορών. Ε, αναφέρεται εδώ πέρα ότι τηρούνται οι προθεσμίες. Παραπληροφόρηση είναι αυτό. Δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση στην Καρόνια. Έχουμε αυτή την επιχείρηση που εκμεταλλευόταν τον πυρηνικό σταθμό. Υποτίθεται ότι σεβόμαστε τη Euratom. Μιλάμε για μια ε, επιχείρηση η οποία δημιούργησε ένα πυρηνικό σταθμό. Το θέμα είναι εκμεταλλεύεται η επιχείρηση το σταθμό αυτό και πρέπει να, να επιφορτιστεί και με τον παροπλισμό. Εγώ δεν νομίζω λοιπόν ότι γίνεται σεβαστή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν γίνονται σεβαστές οι προθεσμίες, γιατί έχουμε μόνο ε, πέντε δοχεία για πυρηνικά απόβλητα. Αγοράστηκαν πέντε δοχεία και αυτό γιατί το κάνανε, γιατί θέλανε ε, να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να αρχίσει το επόμενο εξάμεινο ο παροπλισμός του πυρηνικού σταθμού της Γκαρόνια. Γιατί δεν μπορούν να βγάλουν τα κάψιμα από τον αντιδραστήρα. Δεν έχουν τα δοχεία για να βάλουν τα πυρηνικά, να αποθέσουν τα πυρηνικά κατάλοιπα. Νομίζω ότι σας λείπει πάρα, πάρα πληροφορίες και πραγματικά είναι κρίμα που κλείνεται αυτή την αναφορά. Ευχαριστούμε πολύ. Μα έχει ληφθεί όμω ήδη η απόφαση. Αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να σας στείλουμε τις πληροφορίες παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις Ισπανικές Αρχές και αν στο μέλλον σας δοθεί εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά, τότε έχετε δικαίωμα προφανώς να επαναλάβετε εκ νέου την αφορά σας. Αυτό να αναφέρετε το δικαίωμά σας. Κλείνουμε πάντως αυτή την αναφορά διαδικαστικό πρόεδρο. Please. Yeah, yeah. Point of order is possible. Sí. Eh, pido que por favor se compruebe si hay el... Θέλω να τσεκάρετε καταρχάς την απαρτία, αν υπάρχει επαρκής απαρτία, για να ψηφίσουμε για το κατά πόσον κλείνει αναφορά ή όχι. This is a higher level than the level of the coordinators. Pero quizá no haya quórum en Αν δεν υπάρχει απαρτία στην Επιτροπή, δεν μπορεί να κλείσετε την αφορά. Έχετε δικαίωμα να την ανοίξετε την αφορά στο μέλλον. Αλλά τώρα λήφθηκε απόφαση στην Επιτροπή Αναφορών για να κλείσει η αναφορά. Δεν υπάρχει απαρτία για να ψηφίσουμε αν θα κλείσουμε την αναφορά, καταλαβαίνετε. Πρέπει να ψηφίσουμε για να δούμε αν υπάρχει απαρτία για να κλείσουμε την αναφορά. Αυτό είναι ο κανόνα. Δεν υπάρχει θέμα απαρτία σε αυτήν την περίπτωση. Είναι διπλάσια η σημασία της ψήφου της δικής μου. 665 ε, Είμαι στην επόμενη αναφορά. την 0665 του 17 και την 0198 του 18. Είναι δύο ισπανικές αναφορές πάλι. Σε ό,τι αφορά την μόλυνση του Παλομάρες στην Ισπανία. Είναι εδώ ο αναφέροντας, ο Χωσέ Γνάσιο Μαρτίνες Σάντσες. Έτσι μου είπανε. Είναι εδώ, είναι παρόν. Α, έχετε το λόγο για πέντε λεφτά. Καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ. Θα συνοψίσω το τι συνέβη στο Παλομάρες το 1966. Δύο ε, πολεμικά αεροπλάνα αμερικάνικα συγκρούστηκαν ε, με ένα ε, αεροπλάνο δεξαμενή και κλήθηκαν 9 κιλά πλουτόνιου στην περιοχή αυτή. Έγινε μια εικονική, ένας εικονικός καθαρισμός και οι Αμερικανοί πήραν πίσω στην Αμερική 270 γραμμάρια πλουτόνιου. Τα υπόλοιπα κιλά παρέμειναν στην περιοχή. Υποτίθεται καθάρισαν. Τι κάνανε λοιπόν στην περιοχή. Κάλυψαν το πλουτόνιο το οποίο είχε εξαπλωθεί σε διάφορα ε, χιλιόμετρα με χώμα. Έριξαν από πάνω 20 εκατοστά χώματος σε μια, τριά, ε, σε μια τεράστια έκταση. Επίσης, φτιάξαν και δύο, τεράστια, ε, δύο τεράστιες τάφρους, ε, πηγάδια, ας πούμε, και εκεί θάψανε, ας πούμε, ραδιενεργό υλικό και πλουτόνιο. Έφτιαξαν ένα άλλο πηγάδι, χίλια κυβικά μέτρα, και εκεί θάψανε ραδιενεργό υλικό. Υπάρχει πολύ θόρυβος, νομίζω. Υπάρχουν ακόμα αυτά τα πηγάδια. Είναι ένα νεκροταφείο πυρηνικό ε, παράνομο και στην πραγματικότητα, εκτό από αυτό, τι κάνανε. Καλλιεργούσαν σε προκυπευτικά τα οποία τα εξάγουν σε όλη την Ευρώπη. Η κυβέρνηση του Φράγκο τότε συμφώνησε με τι ΗΠΑ να εξαπατήσει την κοινή γνώμη και τον πληθυσμό του Παλωμάρε, λέγοντα ότι δεν υπήρχε ίχνος ραδιενεργού υλικού. Ενώ ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι είχαν θάψει ε, κάτω από 20 εκατοστά ή σε αυτά τα πηγάδια και τις τάφρους ή σε ζώνες ας πούμε, που δεν, με τις οποίες δεν ασχολήθηκαν πλουτόνιο και το οποίο έμεινε εκεί από το 66. Χάρη στον άνεμο, χάρη στο νερό κτλ. Ε, υπήρχαν ε, άτομα τα οποία ε, περπατούσαν εκεί πέρα, παίρνανε, κάνανε τις βόλτες τους και ανέπνεαν πλουτόνιο. Η φραγκική κυβέρνηση και η αμερικάνικη κυβέρνηση σχεδίασαν λοιπόν να το εξή, να χρησιμοποιήσουν τους α, κατοίκους του Παλωμάρες σαν πειραματόζωα για να δούνε τις επιπτώσεις έχει το πλουτόνιο στην βιολογική ύλη, πάνω στους ανθρώπους, πάνω στο, στην άγρια πανίδα και κλωρίδα, πάνω στο, στα ζώα και στο ε, περιβάλλον. Αυτό έγινε μέχρι το 2003. Κάναν πειράματα με ζώντες ανθρώπους. Οι γεωργοί και οι ιδιοκτήτες των γεών αυτών θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε καθόλου πλουτόνιο στην περιοχή. Κάναν τη δουλειά τους, κάναν τις γεωργικές δραστηριότητες και αυτό το πλουτόνιο κάτω από τα 20 εκατοστά ε, στην πραγματικότητα το ανακάτευαν ας πούμε και δημιουργούνταν ε, ε, ραδιενεργό νέφος ενώ οι Οργανισμό Πυρηνική Ενέργειας και η σημερινή CMAT απλώς σημείωνε τι ραδιενεργή δραστηριότητα είχαμε στην περιοχή και κάνανε μελέτες, μελέτες που υπάρχουν, που δημοσιεύτηκαν για τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας ε, στους ανθρώπους λόγω γεωργικών εργασιών, λόγω κανονική ζωής κτλ. Και μάλιστα κάναμε και συγκρίσει με το Τσερνομπίλ. Στο Τσερνομπίλ Μάλιστα, πρέπει να σα πω, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε του ανθρώπου ω πειραματόζωα. Στο Τσερνομπίλ δεν κάναμε. Ε, δεν δημιουργήσαμε πούμε, ζωντανά εργαστήρια με ανθρώπου. Ενώ στο Παλωμάρε κάναμε τέτοιο εργαστήρι. Με πειραματόζωα ανθρώπου. Και μελέτε. Μάλιστα, όλα αυτά γινόντουσαν μέχρι το 2003. Και από το 2003 και μετά, όχι για ηθικού λόγου, καθαρι... Ε, αποφάσισαν να καθαρίσουν την περιοχή. Για ποιου λόγου αποφάσισαν να καθαρίσουν, Ξεκίνησαν λοιπόν να καθαρίσουν, γιατί δημιουργήθηκε τότε η περίφημη ε, φούσκα των ακινήτων. Θεώρησαν ότι αυτά τα εδάφη είναι εδάφια που μπορούν να οικοδομήσουν, είναι οικοδομήσιμα. Θέλαν να εκμεταλλευτούν λοιπόν τα, τις περιοχές αυτές, άρα να καθαρίσουν ε, από το πλουτόνιο την περιοχή. Ε, αυτό, τον ένα, το ένα πηγάδι λοιπόν με τα χίλια κυβικά μέτρα θα να το καθαρίσουν από το πλουτόνιο. Το 2003 άρχισαν να φτιάχνουν ένα σχέδιο ε, και το 2010 το ε, Συμβούλιο Πυρηνικής Ασφάλειας ε, ένα καταπληκτικό σχέδιο καθαρισμού, το οποίο ήθελε να καθαρίσουν 50.000 κυβικά μέτρα και να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. τελικά όμως αποφάσισαν μετά από διαπραγματεύσεις να μειώσουν αυτό το, αυτό το, το νούμερο σε 28.000 κυβικά μέτρα. Το ανέκρινε αυτό το Συμβούλιο Πυρηνική Ασφάλεια, το είδε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 2010 έστειλε τεχνικού ε, και το είχε δει αυτό το σχέδιο. Τι συνέβη λοιπόν. Το Υπουργείο Ενέργεια των Αμερικανών είπαν, είπε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο και δεν μπορούσε να αποθηκεύσει τόσα πολλά ένα τέτοιο νόγκο. Και πίεσε λοιπόν του Ισπανού. Ε, υπάρχουν έγγραφα μυστικά τα οποία λένε ότι αντί να ε, καθαρίσουμε τα 50.000 κυβικά μέτρα, θα καθαρίσουμε τελικά μόνο τα 28.000 κυβικά μέτρα. Αυτό το σχέδιο το 2015 το ενέκρινε το Συμβούλιο Πυρηνική Ασφάλεια ε, και με την σύμφωνη γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν καταφέραμε το εξή, το οργανισμό να ε, εγκρίνει το καθαρισμό των 28.000 κυβικών μέτρων, συμφωνήθηκε ε, μία συμφωνία μεταξύ του Ισπανικού κράτους και του Υπουργείου Ενέργειας της ε, Αμερικής. Αυτή η συμφωνία όμως όχι μόνο δεν θα, γίνει, δεν θα εφαρμοστεί, Γιατί αντί να καθαρίσουν τα 28 τέλος πάντα χιλιάδες ε, κυβικά μέτρα, στην πραγματικότητα θα συνεχίσουν ε, με το πλουτόνιο, να αφήνουν το πλουτόνιο στην περιοχή. λοιπόν στην ουσία παραβιάζεται η οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια και ο νόμος και σε εθνικό και σε, κοινωνικό, και σε κοινοτικό επίπεδο. Ο Χωσέ έχει το λόγο. Buenas Επί 53 χρόνια στο Παλομάρες ζούμε με την ραδιενέργεια. Στην ουσία είμαστε 25 χιλιόμετρα από ε, <clears throat> το σημείο από το οποίο προέρχεται η αναφορά. Από τις έξι ζώνες που έχουν μολυνθεί ραδιενεργά, οι πέντε είναι γύρω από την ε, περιφέρεια της συγκεκριμένης Χερσονήσου. Ξέρετε ότι το ατύχημα στο Παλωμάρες ε, ήταν στον ψυχρό πόλεμο. Υπήρχαν 10 κιλά πυρηνικού καυσίμου στην βόμβα η οποία έπεσε κατά λάθο. 20 χρόνια μετά στο Τσερνομπίλ θεωρήθηκε το πιο σημαντικό ατύχημα της πυρηνικής εποχής. Θυμίζουμε εδώ ότι ήταν η πρώτη φορά ...που μία βόμβα υδρογόνου στη συγκεκριμένη περίπτωση έπεσε ε, πάνω σε πληθυσμό εκτός Χειροσύμα και εκτός ε, ε, Ναγκασάκη. Βλέπουμε εδώ τη ζώνη 0, όπως καθορίστηκε το 1966 υπήρξε μια ηγετικού τύπου συμπεριφορά πάνω σε μια χώρα η οποία ήταν υπηρέτης και την οποία διοικούσε μια δικτατορία. Βλέπουμε σε κλίμακα μια, έναν χάρτη ότι στην ουσία έχει υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια μόλυνσης και υπάρχουν επίσης και περιοχές οι οποίες ε, δεν έχουν συμπεριληφθεί και δεν περιλαμβάνονται και στις φωτογραφίες της ζώνης της που έχει μολυνθεί. Από το 2000 υποτίθεται ότι υπάρχει μια δυνατότητα διαγενειακής καταμέτρησης σε σχέση με την ε, διεύρυνση της ζώνης του Παλομάρες. Υπάρχει, ε, θα έλεγα, επέκταση της ζώνης μέσα στις οποίες κινούνται οι κάτοικοι υπάρχει ένα κριτήριο ραδιολογικό, ραδιολογικού τύπου το οποίο ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια μιας μελλοντικής προσπάθειας ε, από ε, ραδιενεργοποίησης στην ουσία. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο σε καμία περίπτωση δεν φτάνει σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η μείωση κατέτος είναι πάρα πολύ χαμηλή, ελάχιστη και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ελεγχθεί και από την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 5 της ΕΡΑΤΟΜ σχετικά με τη ζώνη αποκατάστασης. Στις νέες μελέτες οι οποίες έγιναν, φέρεται ότι ε, ο κατάλογος των σημείων που δεν περιλαμβάνονται έτσι και αλλιώς πλήρως στις αμερικανικές μελέτες και έτσι και αλλιώς έχουν ε, τα στοιχεία αυτά αλλοιωθεί από τις πλημμύρες που κατά καιρούς έχουν χτυπήσει την περιοχή, αλλά μόνο από το 2008 έχει υπάρξει πλήρης απαγόρευση χρήσης. 50 χρόνια ο κόσμος ζούσε εκεί, καλλιεργούσε εκεί, φύτευε εκεί και δεν υπήρχε ουσιαστική προειδοποίηση και βλέπετε ακριβώς και μία ζώνη στο κέντρο ακριβώς αυτής της ζώνης, της πόλης, ε, στη ζώνη 3. Η ζώνη αυτή λοιπόν περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Κέρι Μαργκάγιο, τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών δηλαδή, στην ουσία περιλαμβάνεται καταγραφή ενός μπεκερέλ Sin embargo, en la του Αμερικίου 241. Στην ουσία όμως απεδείχθη ότι ε, έχουμε τώρα τέσσερα μπέκερελ αναγραμμάριο ε, της ουσίας αυτής, ε, δηλαδή 400% ουσιαστικά περισσότερο και με αυτό φύγει μια περιοχή η οποία έχει θα έλεγα τουριστικό μέλλον εξαιρετικό, έχει μια εξαιρετική παραλία και αυτά όλα καθυστερούν λόγω της ηγεμονικής τάσης της συγκεκριμένης χώρας Στην ουσία η συγκεκριμένη χώρα δεν είχε κανένα πρόβλημα το 2015 και υποβίβασε ουσιαστικά τις απαιτήσει του και τα κριτήριά του και ενέκρινε την Αμερικανική πρόταση. Υπάρχουν λοιπόν, έχει αποφασιστεί κάποιες επιμέρου μορφές περιορισμού στο μέλλον, γιατί η λήψη στοιχείων δείχνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει αύξηση της παρουσίας Αμερικίου. Αυτό σημαίνει ότι για μια ακόμη φορά γίνονται τα ίδια πράγματα και το τίμημα, το κοινωνικό και κυρίως το οικονομικό που έχουμε πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια θα παραταθεί για 400 τόσα χρόνια, κάτι το οποίο είναι ο χρόνος τον οποίο ε, θα χρειαστεί να διανύσει ώσπου να εξαφανιστεί συγκεκριμένη ουσία και αυτά όλα με τέσσερις περιοχές οι οποίες ε, θα περιοριστούν πλέον και με πολλές βλάβες για τον τουρισμό και την οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω πάλι το λόγο στην κυρία Σέικα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε πάλι το λόγο να ευχαριστήσω του αναφέροντες για πολύ ενδιαφέρουσες και εξαντλητικές παρουσιάσεις στο θέμα του Παλωμάρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα καταρχάς να τονίσει ότι καταλαβαίνει πολύ καλά τις ανησυχίες των Ισπανών πολιτών για το Παλωμάρες και συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση ε, στο θέμα αυτό. Όσον αφορά το αίτημα να πραγματοποιηθεί διαρευνητική επίσκεψη στο Παλωμάρε, έχουμε το άρθρο 35 που μπορεί να αποτελέσει βάση μιας τέτοια αποστολή. Ε, και με χαρά σας ενημερώνω ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίσκεψη στο πρώτο εξάμεινο του φετινού έτους ε, και θα εξεταστεί και η εφαρμογή των συστάσεων που ε, εστάλησαν μετά την προηγούμενη ε, αποστολή. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η Ισπανία και, και οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία για το, την αποκατάσταση του Παλωμάρες ε, που αναφέρθηκε του 2015. Και οι δύο κυβερνήσεις εξέφρασαν την πολιτική τους βούληση να συνεργαστούν για την αποκατάσταση της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης ε, της ε, μεταφοράς των αποβλήτων και την τελική τους αποθήκευση στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ως αποτέλεσμα, εκκρεμεί ακόμη και η τελική έγκριση του σχεδίου αποκατάστασης του Παλωμάρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας υποβάλει έκθεση σχετικά με την επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 της συνθήκης. Αυτό που να το περιμένετε το δεύτερο εξάμεινο του φετινού έτους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευρωβουλευτές, η κυρία Αλπιόλ. Σας ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν έχουμε πολλά να συζητήσουμε και στο τέλος θα λυθεί το θέμα με μία ψηφοφορία. Είμαστε έξι βουλευτές εδώ, ε, τρεις πολιτικές ομάδες ε, και χωρίς να έχουμε το απαιτούμενο, την απαιτούμενη απαρτία. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι απαράδεκτη, ε, δεν έχει ξαναγίνει. Θέλω να ευχαριστήσω, εν περιπτώσει, αυτούς οι οποίοι κατέθεσαν την αναφορά. Είναι σαφές ότι η δήλωση του 2015 σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανοποιητική και δεν περιλαμβάνει την επιθυμία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και οι Ισπανικές αρχές και οι Ευρωπαϊκές αρχές στην ουσία δεν βοήθησαν τον πληθυσμό, ο οποίος πληθυσμός εδώ και 15 χρόνια περιμένει τον καθαρισμό la población local, lo cual es sin ε, νομίζω ότι αυτό επηρεάζει αρνητικά φυσικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής όπως και το δικαίωμα ενημέρωσης του πληθυσμού. Πρέπει να παραμείνει συνεπώς λοιπόν η αναφορά ανοιχτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει με την προσπάθεια την οποία έχει ξεκινήσει για τον έλεγχο της κατάστασης. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπε η Επιτροπή για την αποστολή το πρώτο τρίμηνο του 2019. Εμείς θα περιμέναμε περισσότερα στοιχεία. Πότε ακριβώς θα γίνει δηλαδή η συγκεκριμένη αποστολή. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει το άρθρο 75 ε, της συνθήκης Ερατόμ και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα περισσότερο χρόνο έτσι ώστε να ε, επιληθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ε, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να πετύσει από την Ισπανική κυβέρνηση ένα λεπτομερές πρόγραμμα και με πολύ συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να περάσουμε τη διαδικασία απομόλυνσης της περιοχής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους αναφέροντες που ήρθαν ως εδώ για να μας μιλήσουν και να μας μεταφέρουν την άποψή τους για ένα σκάνδαλο υγειονομικό, σκάνδαλο πυρηνικής μόλυνσης και γεωπολιτικό σκάνδαλο. Έτσι, πρέπει να το δούμε με σαφήνεια από όλες τις απόψεις. Ε, αυτά που μας υποσχέθηκαν δεν έγιναν, δεν υπάρχει πρόγραμμα σαφές ε, για να αντιμετωπιστεί αυτό το σκάνδαλο σε αυτή τη φάση. Στηρίζω αυτή την αναφορά των κατοίκων του Παλωμάρες, μετά από 53 χρόνια που παραμένει το πρόβλημα, νομίζω ότι για, σεβασμό, για σεβασμού απέναντι στους κατοίκους πρέπει τουλάχιστον να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πάει επί τόπου για να διαπιστώσει τι έχει γίνει και να ληφθεί μια απόφαση πραγματική. Γιατί όλοι γνωρίζουμε τη σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζει το Παλωμάρες. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ένα διαδικαστικό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη με την προηγούμενη ψηφοφορία, την οποία δεν θεωρώ έγκυρη, γιατί οι κανόνες είναι σαφείς. Ε, ο, το άρθρο 178 ε, και το άρθρο 229 λέει ότι πρέπει να έχουμε απαρτία για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Το 1 τρίτο για τους 10 ε, είμαστε 6, δεν έχουμε απαρτία. Ε, πρέπει να δούμε και τις ε, κατευθύνες γραμμές της Επιτροπής ΠΕΤΗ του 2015 και λέει ότι αν δεν υπάρχει απαρτία, ε, το θέμα θα πρέπει να το να φορτιστεί με το θέμα αυτό οι συντονιστέ. Εκεί πρέπει να πάει το θέμα, στους συντονιστέ. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Μόνο αν υπάρχει συνένεση με βάση του κανόνε. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω από τον Πρόεδρο να σεβαστεί του κανόνε του οίκου μα. Σα ευχαριστώ πολύ. θα παρακαλούσα τη Γραμματεία να μεταφέρει αυτή την απόφαση στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών. Συμφωνείτε? Ωραία. Και συνεχίζουμε τη συζήτηση. Κύριε Χιμένες, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους αναφέροντες που ήρθαν εδώ. Δεν γνωρίζω με λεπτομέρειες τα συμβάντα στο Παλεμάρες, αλλά είναι λίγα τα άτομα στην Ισπανία που δεν γνωρίζουν πόσο σοβαρό είναι αυτό το ατύχημα. Ειδικά οι πιο μεγάλοι στην ηλικία από εμά θυμόμαστε το ατύχημα. Γιατί η Αλμερία είναι στην Ανταλουσία έτσι, και το Παλομάρες είναι στην Ανταλουσία και ήταν σαφή σε όλους μας στην ε, Ανταλουσία ότι υπήρχε κίνδυνος και όπως πολύ σωστά είπαν οι αναφέροντες, καμία από τις κυβερνήσεις που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε τίποτα. Ούτε σε κρατικό επίπεδο έγινε τίποτα, ούτε σε περιφερειακό επίπεδο έγινε τίποτα. Οι περιφερειακές κυβερνήσεις δεν έλαβαν υπόψη τους ότι πρόκειται για την ζωή, την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ε, να παίρνουν αποφάσεις για τη γεωργία και τα λοιπά, χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος. Στηρίζω λοιπόν την ιδέα για την επίσκεψη επιτόπου. Πρέπει να γίνει μια τέτοια επίσκεψη για να διευκρινίσουμε τις, τα συμβάντα και για να ανασάνει λιγάκι ο πληθυσμός. Γιατί ζουν όλα αυτά τα χρόνια σε μια περιοχή που είναι μολυσμένη από ραδιενέργεια. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει συνένεση γύρω από αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει στη ζωή του Παλωμάρες. Έχει στιγματιστεί η περιοχή αυτή και σε τομείς όπως η γεωργία, όπως και ο τουρισμός και θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους ομιλητές. Κοιτάξτε, ε, στην δημοκρατία πάντα υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο κάνει κάποιους να κερδίζουν και άλλους όχι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε την υποχρέωση να είμαστε εδώ, αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε παρόντες, αλλά εδώ λείπουν οι μισές πολιτικές ομάδες αλλά δεν θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ασέβεια απέναντι στους αναφερόμενους από πλευράς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ε, ο σεβασμός οφείλεται στους παρόντες. Αυτό έχει σημασία. Πρέπει κανείς να είναι παρόν. Αυτή είναι η δημοκρατία, τον σεβασμό στους αναφερομένους τον δείχνουμε εμείς που είμαστε παρόντες και παρούσες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι προφανές το τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να περιμένουμε τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και τα αποτελέσματα της αποστολής. Προφανώς αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί η επόμενη θητεία. Διότι τα συμπεράσματα θα εξαχθούν το δεύτερο εξάμεινο του έτους. Ελπίζουμε λοιπόν το μελλοντικό κοινοβούλιο να ασχοληθεί με αυτό και να είναι περισσότεροι ευρωβουλευτές παρόντες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται να υπάρχει συνένεση λοιπόν. Θα διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της ε, διαρευνητικής επίσκεψης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύο λεπτά έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ για τη στήριξη στην ε, αναφορά μας. Θα ήθελα να πω το εξής. Αυτό που προτείνουμε εμείς, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε δικαστικό επίπεδο, γιατί πήγαμε στο το δικαστήριο της Ισπανίας, είναι να μην τηρηθεί η συμφωνία με τους Αμερικανούς και να αυτά τα 50.000 κυβικά μέτρα να αποθηκευθούν προσωρινά. Αυτή τη στιγμή βρούμε προσωρινή αποθήκη να κάνουμε διαπραγματεύσει ε, ξανά με του Αμερικανού μέχρι να βρούμε πραγματικό και οριστικό νεκροταφείο. Δηλαδή, καταρχά να καθαρίσουμε, να αποθυματοποιήσουμε προσωρινά και εν συνεχεία να διαπραγματευτούμε για την οριστική αποθυματοποίηση. Θα ήθελα επίση να πω ότι υπάρχει μια φοβερή μυστικοπάθεια γύρω από αυτά. Γιατί το σχέδιο που υπερασπιζόμαστε ε, και μάλιστα εγώ ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου ε, μίλησα για το σχέδιο του 2010 που ήταν μυστικό στο ανώτατο δικαστήριο δεν μου δίνουν το έγγραφο που έστειλαν οι Αμερικανοί, γιατί είναι μυστικό για να μάθω την πραγματικότητα. Επίσης, η συμφωνία του 2015 είναι μυστική. Εμείς στο Παλωμάρι, λοιπόν, ζούμε ε, από αποχαρακτηρισμό σε αποχαρακτηρισμό εγγράφου που γίνονται περιοδικά, ας πούμε, και ε, παρακολουθούμε τι δημόσιε δηλώσει που κάνουν οι διάφοροι αξιωματούχοι, α πούμε. Θα τελειώσω, έτσι. Είναι τεράστια σοβαρότητα του συμβάντος. Τα παιδιά κυκλοφορούν στους δρόμους. Υπάρχουν 62.000 ε, μπεκερέλ του Αμερικίου 241 που εισπνέουν τα παιδιά όταν κυκλοφορούν και κάνουν τη βόλτα τους ή παίζουν στους δρόμους. Ένα λεπτό από μένα. Από το 1966, κάθε φορά που διαβάζω ένα άρθρο, το άρθρο 35 μάλλον της συνθήκης ε, Euratom, ε, σκέφτομαι ότι ποτέ δεν τηρήθηκε αυτό το άρθρο. Γιατί αν, ήμασταν, αν το είχαμε τηρήσει, δεν θα είχαμε φτάσει εκεί που φτάσαμε με αυτό το ραδιολογικό κατάλογο που φτιάχνουμε. Το θέμα δεν είναι να πάει μια επιτροπή διερευνητική ε, επιτόπου. Το βασικό, το βασικό θέμα, ο βασικός στόχος είναι να γίνει καθαρισμός του, της περιοχής. Ε, με ή χωρίς τους Αμερικάνους. Πέρασαν 53 χρόνια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ε, τα, τις αποφάσεις πολύ μακριά από μας και η προτεραιότητά τους δεν είναι η καθαρότητα του ισπανικού περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην αναφορά 327 του 2018 που έχει να κάνει με την εγκατάσταση διάθεσης πυρηνικών αποβλήτων Ελκαβρίλ στην Κόρδοβα. Αναφέρον είναι ο Σεμπαστιάν Πέρες Χαλιάρδο. Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών ε, ήδη κατετέθη τις 18 Ιουλίου του 2018. Αναφερόμαστε στο λεγόμενο πυρηνικό νεκροταφείο του Γαβρίλ. Πρέπει να δούμε πώς έχει η κατάσταση, όπως ε, δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο ελέγχεται σε σχέση με την πιθανή όχληση που μπορεί να προκαλέσει προς τον πληθυσμό. Εγώ είμαι εκπρόσωπος ε, των πληθυσμών που θίγεται στην περιοχή σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο εκπροσωπούνται στα πλαίσια αυτής της αναφοράς πάρα πολλές οργανώσεις, πολιτικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κτλ. κτλ. Εμείς θεωρούμε το εξής εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το πρόβλημα ακριβώς της, πυρηνικής, της πυρηνικής ενέργειας, της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας είναι η διάρκεια ζωής του υλικού το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, του καυσίμου το οποίο έχει ήδη ε, χρησιμοποιηθεί και το οποίο είναι, εκπέμπει σε ε, χαμηλή ε, ή μεσαίου τύπου εκπομπές ραδιενεργές η αντιμετώπιση, η διαχείριση αυτών των ε, πυρηνικών αποβλήτων δεν έχει υπολογιστεί ακριβώς τι ζημίες μπορεί να προκαλέσουν σε επίπεδο κοινωνικό, σε επίπεδο επίσης ιατρικό. Δεν μπορούμε να πούμε όμως το ίδιο ότι ε, τα απόβλητα ε, χαμηλής... Como los de alta. Sin embargo, no Τα κάψιμα λοιπόν τα πυρηνικά τα οποία έχουν συμμετοποιηθεί και είναι πλέον α, ε, α, έχουν αναλωθεί μέχρι τώρα έχουν αποθηκευθεί στο λεγόμενο πυρηνικό νεκροτραφείο του Γαβρίλ στην Ανδαλουσία υποτίθεται ότι έχουν περιορισμένη δραστηριότητα, έχουν μία μεσαία διάρκεια ζωής γύρω στα 30 χρόνια και δεν εκπέμπουν υψηλή δραδιενέργεια ε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν γίνονται σεβαστοί οι κανόνες από την συγκεκριμένη επιχείρηση διαχείρισης. Η δημόσια επιχείρηση, η ΕΝΡΕΣΑ, ε, είναι υπεύθυνη για την ε, διαχείριση των αποβλήτων. Έτσι κι αλλιώς ε, η ηγεσία αυτών των δομών έχει εκλεγεί με μη δημοκρατικό τρόπο και τα πρώτα πυρηνικά απόβλητα ήρθαν το 71 στην περιοχή, προέρχονται από από ε, τον στρατό έχουν κληρονομηθεί στον Ισπανικό στρατό από ε, τους Αμερικανούς δόθηκε μία μάχη νομική ε, η οποία κερδίθηκε το 2002. Υπήρξε έτσι κι αλλιώς απόφαση του Ανωτάτου Δικητικού Δικαστηρίου της Μαδρίτης υπέρ ημών Η απόφαση αυτή αναγνωρίζει ότι η εναπόθεση των αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας διενέργειας ήταν παράνομη. αλλά υπήρξε στην ουσία εν τω μεταξύ μια διεύρυνση της περιοχής του Γαβρίλ, στην ουσία οικοσαπλασιάστηκε η χωρητικότητά του. Υπάρχει, είναι σαφής η έλλειψη εμπιστοσύνης, η έλλειψη διαφάνειας, η έλλειψη ε, εμπιστοσύνης. Είναι προβληματική η τοποθέτηση στο Καβρίλ γιατί στην ουσία υποδέχεται ε, τα απόβλητα όλων των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Επίσης είναι πάρα πολύ κοντά σε ένα τοπίο το οποίο είναι υψηλής, ε, υψηλού φυσικού κάλους και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ασφαλείας. Δεν εκτιμάται ο κίνδυνος ο οποίος δημιουργείται από τα απόβλητα αυτά με αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Και επίσης η μεταφορά των υλικών των πυρηνικών έχει προκαλέσει και ατυχήματα. Υπάρχουν δύο δηλωμένα ατυχήματα και μάλιστα στα πλαίσια του ενός χρειάστηκε να υπάρξει απομόλυνση του εδάφους πάνω στο οποίο έγινε το ατύχημα. Υπήρξαν επίσης ε, και ε, πυρκαγιές που απέδειξαν ότι τα συστήματα αντιμετώπισης της φωτιάς της πυρκαγιάς ε, δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Και μάλιστα πιο πρόσφατα υπήρξε άνοδος ε, του ε, η διαχείριση, εν πάση περιπτώσει, των υδάτων από τις βροχές δεν μπόρεσε να γίνει σωστά αντικείμενο αντιμετώπισης. Είναι προφανές ότι θα χρησιμοποιηθεί, προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο ε, ε, μετά την ε, πάυση λειτουργίας της πυρηνικής μονάδας η οποία βρίσκεται, το παροπλισμό πυρηνικών παλαιών μονάδων Λοιπόν δεν υπάρχει κανένας οικονομικός ή περιβαλλοντικός λόγος που θα επέτρεπε ε, ε, να ενισχυθεί ο χώρος αυτός, ο οποίος έχει προκαλέσει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και περιβαλλοντικά προβλήματα. Υπάρχει κοινωνική συνένεση για να βρεθεί ε, ένας χώρος εναποθήκευσης του υλικού αυτού χαμηλής και μεσαίας εκπομπής ραδιενέργειας Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι από τη μεταφορά του υλικού, δεν λαμβάνεται επίσης υπόψη η σεισμική ασφάλεια της περιοχής και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση στην, στην ισπανική κοινωνία όπως επίσης ε, μια συζήτηση και σε ευρωπαϊκό, όχι μόνο σε ισπανικό επίπεδο, για τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας που να είναι ασφαλείς και καθαρές. Θα πρέπει να υπάρξει, λοιπόν, απαιτούμε να υπάρξει μια αποστολή στο Καβρίλ από ευρωβουλευτές και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφασή της να επισκεφτεί άλλες περιοχές. Οι ε, Ισπανικές αρχές παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε σχέση με την υποχρέωση ενημέρωσης και σε σχέση με την διαφάνεια και την επικινδυνότητα του προγράμματος στην περιοχή υπάρχει έλλειψη και σε επίπεδο ενημέρωσης και σε επίπεδο τεκμηρίωσης, όπως επίσης και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από την μονάδα παραγωγής Σαντα Μαρία του ε, Δεκαρόνια από τον Μπούργος, τα οποία απόβλητα αυτά είναι υψηλής ε, ε, εκπομπής ραδιενέργειας. Παραβιάζονται οι κανόνες λοιπόν για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, εναποθηκεύονται ε, απόβλητα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην άδεια λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας, όπως επίσης και ε, ουράνιο ε, το οποίο προέρχεται από την μονάδα παραγωγής της Σαλαμάνκα και παραβιάζεται πλήρως το αντίστοιχο άρθρο της συνθήκης ε, Ερατόμων. Θα κλείσω την παρέμβασή μου εδώ ζητώντας ε, να υπάρξει ε, παρέμβαση η οποία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο τοπικός πληθυσμός, να επαληθευτεί το είδος των αποβλήτων τα οποία αποθηκεύονται στο Καβρίλ, και να υπάρξει επιτέλους μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που να λάβει υπόψη τις ε, συνέπειες της αποθήκης αυτής πυρηνικών αποβλήτων στην φυσική ζώνη που περιβάλλει το χώρο. Uh, thank you very Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Καγιάρτο. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα για άλλη μια φορά να πει ότι καταλαβαίνει πολύ καλά τις ανησυχίες σας. Καταλαβαίνουμε ότι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ανησυχούν σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων πυρηνικών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, διέπεται από την οδηγία περί αποβλήτων και υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ε, ένα ε, σχετικό ε, νομοθετικό και αριθμιστικό πλαίσιο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την συμμόρφωση με την οδηγία και να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της. Ειδικά αυτή η οδηγία ζητάει από κάθε κράτος μέλος να δημιουργήσει ένα εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση χρησιμοποιημένων καυσίμων και πυρηνικών αποβλήτων και να υποβάλει σχετικές εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει τέτοιο πρόγραμμα από τις Ισπανικές Αρχές ε, που συμπεριλαμβάνει και τη δημιουργία πρόσθετης εγκατάστασης για τη, τα πυρηνικά απόβλητα του El Cabril για την διαχείριση αποβλήτων ε, πυρηνικών χαμηλού κινδύνου. Το 2018 επιπλέον οι Ισπανικές αρχές υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας. Η έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το είδος πυρηνικών αποβλήτων που αυτή τη στιγμή ε, ε, τοποθετούνται στην εγκατάσταση El Capril. Επίσης συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις ε, για τη μελλοντική χρήση της εγκατάστασης δεν έχει δηλωθεί ε, να ε, υπάρχουν ε, πυρηνικά αποβλητά υψηλού κινδύνου στο El Καμπρίλ. Ωστόσο, η τελική ευθύνη για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων ανήκει στα κράτη-μέλη που παράγουν τα απόβλητα αυτά, το οποίο σημαίνει ότι οι Ισπανικές Εθνικές Αρχές είναι υπεύθυνε για την μεταφορά πυρηνικών αποβλήτων στο El Καμπρίλ. και για τη συμμόρφωση με τις ε, εθνικές ρυθμίσεις για την ε, ασφαλή και υπεύθυνη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Επιπλέον, η συνθήκη Ευρατόμ απαιτεί από τα κράτη-μέλη να παρακολουθούν τα επίπεδα ραδιενέργειας ε, στον αέρα, τα ύδατα, το έδαφος και τα τρόφιμα και να υποβάλουν τα σχετικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δυνατότητες παρακολούθησης ε, της κατάστασης. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να προσθέσει ότι η κατασκευή και τροποποίηση της εγκατάστασης El Cabril ε, έγινε κατόπιν ε, κανονικής μελέτης αντικτύπου και οι Ισπανικές αρχές κατέληξαν ότι η δημιουργία αυτής της εγκατάστασης δεν ε, θα είναι εις βάρος ε, των περιοχών Natura 2000. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέρφους μου, αν θέλει κανείς το λόγο. Κύριε Αλβιόλ, παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ. Βλέπω ότι σε αυτή την αναφορά για την οποία θέλω να ευχαριστήσω τους αναφέροντες, υπάρχουν λοιπόν τρία ουσιαστικά στοιχεία. Καταρχάς, ο πληθυσμός απορρίπτει τις εγκαταστάσεις αυτές. Δεύτερον, οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται σε μία ζώνη που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 υψηλής προστιθέμενης αξίας, ε, με σεισμική σεισμογενή δραστηριότητα, δεν τηρείται η αρχή της πρόληψης και δεν υπάρχουν πληροφορίες, δεν υπάρχει διαφάνεια για το ποιο κατάλοιπα αποθηκεύονται σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Με βάση αυτά τα τρία στοιχεία, νομίζω ότι εμείς ως Επιτροπή Αναφορών πρέπει να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από τις Ισπανικές Αρχές και να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά μέχρι να μας έρθουν αυτές οι πληροφορίες και να μπορέσουμε να τις αναλύσουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Colleague please. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ο Μαρθελέση. Ευχαριστώ τους αναφέροντες ε, και όλες τις οργανώσεις ε, που του στήριξαν και βοήθησαν στο να φτάσει το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πυρηνική ενέργεια είναι ένας κλάδος οικονομικός ε, που διέπεται από αδιαφάνεια δεν υπάρχουν αρκετέ πληροφορίε και βλέπουμε και με αυτή την περίπτωση, αλλά είδαμε και με τι υπόλοιπε περιπτώσει που εξετάσαμε πριν, στην Καρόνια ή στο Παλωμάρε, πόσα προβλήματα διαφάνεια υπάρχουν. Νομίζω ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι, να ζητήσουμε περισσότερε πληροφορίε. Οι πολίτε πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει με την πυρηνική ενέργεια. Δεύτερον, εξακολουθούμε να έχουμε αμφιβολίε παρά τα όσα μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν έχει ακολουθηθεί σωστή διαδικασία και έχουν γίνει σωστέ περιβαλλοντικέ μελέτε αντικτύπου για την περίπτωση του Ελκαμπρίν. Έχουμε σοβαρέ αμφιβολίες, όπω είπαν και οι αναφέροντε, για την ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι το άπαν σε ό,τι αφορά την ε, πυρηνική ενέργεια, δεδομένων των ε, κινδύνων που ενέχει η πυρηνική ενέργεια. Διπλή ασφάλεια. Έχουμε και του σεισμού. έτσι. Όταν μιλάμε για την πυρηνική ενέργεια, η πυρηνική ενέργεια έχει δυνατότητα να καταστρέψει τα πάντα. Και επιπλέον μην ξεχνάτε, ε, όποιο γνωρίζει την Ισπανία, στην πραγματικότητα μεταφέρουμε από τον βορρά στον νότο. Όσο πιο μακριά είναι, τόσο πιο επικίνδυνο είναι. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτού του κινδύνου. Επομένω, με όλα αυτά, νομίζω είναι σημαντικό να μην ανοιχτή η αναφορά. Επίση, θα ήθελα να ξαναδούμε το θέμα της επίσκεψης, όχι μόνο να επισκεφτούμε το El να επισκεφθούμε το σύνολο τη Ισπανία, να δούμε τι διάφορε εγκαταστάσει, να δούμε την κατάσταση που υπάρχει, ε, για να δούμε αν συνολικά σέβεται τι οδηγίε ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ισπανία. Είτε στην Καρόνια, στον Παλωμάρε, στο Ελγκαρίλ, να κάνουμε μια συνολική επίσκεψη με όλε τι πολιτικέ ομάδε με σωστή πληροφόρηση, με απόλυτη διαφάνεια, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Η κυρία Σταράς Φεραγκούτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους αναφερομένους. Άκουσα την Επιτροπή και μπορώ να πω ότι δεν συμφωνούμε στην ουσία. Ε, να δεχθούμε τη λογική της ε, αποθήκευσης ε, των αποβλήτων των πυρηνικών χωρίς να υπάρχει πλήρης κάλυψη σε σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τις κοινοτικέ εγγυήσεις, τις εγγυήσεις ε, από την ε, ραδιενέργεια και τις εγγυήσεις προστασίας ε, από τα απόβλητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι καλύπτονται κάποιες απαιτήσει σε σχέση με την προστασία από τα απόβλητα, ότι με σωστό τρόπο η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν έχει σημασία ποια είναι η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ελέγχεται από την Επιτροπή, ελέγχεται από την Ερατόμ για την ασφάλεια, για τον πληθυσμό, για το περιβάλλον και γενικότερα για τον σεβασμό των κανόνων και οι κανόνες γίνονται σεβαστοί με επακριβέστατο τρόπο. Εγώ είμαι δικηγόρος και ήμουν βουλευτής στις Βαλεαρίδες και καταλαβαίνω τις δυνατότητες που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ φυσικά δεν είμαι εναντίον της περαιτέρω λήψης μέτρων, διότι θα πρέπει να καθησυχάσουμε τον πληθυσμό και να είναι καλύτερα ενημερωμένος αλλά η πληροφόρηση μετά από αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την πρόληψη, την ενημέρωση, την τεκμηρίωση είναι ε, σε ικανοποιητικό επίπεδο και δεν βλέπω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε επιπλέον. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να θέσουμε σε αμφιβολία ε, αυτά τα οποία είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι πολιτικό όργανο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι τεχνικό όργανο Δεν ξέρω αν υπάρχουν επιχειρήματα επιστημονικά τα οποία θα μπορούσαν να διαψεύσουν αυτά τα οποία ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στηρίζω αυτά που είπε η συνάδελφος Ρώσα Εσταράς και άλλοι ευρωβουλευτές και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει διάσταση απόψεων εδώ. Εδώ τι θέλουμε, να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες. Η διαφορά με τις προηγούμενες ε, αναφορές είναι ότι δεν αμφισβητούμε αυτά που μας είπε η Κομισιόν, η οποία έχει αυτή την έκθεση. Ο πληθυσμό όμω ανησυχεί, είναι σαφές. Είναι λογικό να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για να είναι ξεκαθαριστεί το θέμα. Άρα εγώ δεν θα αντιταχθώ στο να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά σε καμία περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται να υπάρχει συνένεση. Θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και θα ζητήσουμε με επιστολή περισσότερα στοιχεία. Κύριε Καγιάρδο, τελε, τελικές παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ για το γεγονός ότι κρατάτε ανοιχτή την αναφορά. Νομίζω είναι σημαντικό. Υπάρχει αδιαφάνεια για το πώς δημιουργήθηκε το Ελκαμπρίλ και το τι συμβαίνει στο Ελκαμπρίλ. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας είναι καταφανής. Νομίζω ότι με παράνομο τρόπο δημιουργήθηκε και συστήθηκε αυτό το Ελγκαρίλ, γιατί υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που λένε κάτι τέτοιο, ότι ήταν παράνομο, παράνομη γέννηση και δημιουργία. Πέρα από το γεγονός ότι κρατάμε ανοιχτή την αναφορά, είναι βασικό να γίνει μια επίσκεψη επιτόπου στο νεκροταφείο αυτό και να γίνει μια πραγματική αξιολόγηση του τι γίνεται. Γιατί μπορούμε να αποδείξουμε ότι πρόσφατα έγιναν ε, ατυχήματα στο Ελκαμπρίλ. Ε, είναι κίνδυνος για τον πληθυσμό, πραγματικός κίνδυνος. Και μην ξεχνάτε ότι οι μεταφορές αυτών των πυρηνικών ε, καταλήπων γίνονται ε, από τους, μέσω των αυτοκινητοδρόμων, έτσι, χερσαίως. Περνάνε από πολλούς δήμους και κοινότητες στη διαδρομή αυτή τα πυρηνικά απόβλητα ε, αν το προσθέσουμε με, τους, ε, με τη σεισμική δραστηριότητα που υπάρχει στην περιοχή, δεν θέλω να μακρηγορήσω πολύ, αλλά θέλω να σας πω ότι σε καμία περίπτωση η επαρχία της Κόρδοβας και ο βορράς ε, της επαρχίας αυτής και η Σεβίλη δεν μπορούν να απτυχθούν με αυτόν τον τρόπο, ούτε κοινωνικά ούτε οικονομικά. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τον Ελκαμπρίλ ε, μειώνεται ο πληθυσμό, δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Χάνουμε τον πληθυσμό μας, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πολύς πληθυσμός φεύγει. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το νεκροταφείο του Ελκαμπρί. Πρέπει να γίνει αυτή η επίσκεψη, είναι απαραίτητη. Είναι σημαντικό να δοθούν οι πληροφορίες από την Ισπανική κυβέρνηση μετά τα ατυχήματα που έγιναν, ε, μετά το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση, θεωρούμε, αμφισβητούμε αυτά που λέει η Ισπανική κυβέρνηση και οι αρχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επαναλάβω την απόφασή μας. Η απόφασή μας είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας διαβιβάσουμε τις πληροφορίες που περιμένουμε. Μάλλον βέβαια η επόμενη, το επόμενο κοινοβούλιο θα αποφασίσει. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε στην αναφορά 14 98. Πρόκειται για αναφορά που έχει να κάνει με ένα πρόβλημα περιβαλλοντικής ρήπανσης. Κύριε Όρος, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε περιβαλλοντικό θέμα. Μιλάμε για τη Σλοβακία. Επιτρέψτε μου σύντομα να σας περιγράψω το πρόβλημα. Η Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της Σλοβακίας, απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την περιφέρεια Βερέκνιε, γνωστή επίσης ως Βράκουνα. Υπάρχει εδώ παραπόταμος του Δούναβη. τη δεκαετία του 80 ή του 90. Αποθηκεύθηκαν πολλά επικίνδυνα απόβλητα στην περιοχή αυτή. Αυτό ήταν παράνομο και αυτό σήμαινε ότι δημιουργήθηκε έτσι μια παράνομη κατάσταση. Μιλάμε για 120 ε, κυβικά μέτρα νερού που έχουν επηρεαστεί από αυτό. Μιλάμε για χημικά προϊόντα, για παραπροϊόντα φυτοφαρμάκων, τα οποία έχουν ταφεί σε ε, βαρέλια κάτω από το έδαφος. Ε, κατά τη διάρκεια των ετών έχουν σκουριάσει και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τα υγρά που περιέχονται σε αυτά τα βαρέλια είναι επικίνδυνα χημικά και σιγά σιγά διαραίουν ε, στον υδροφόρο ορίζοντα. Πρόκειται για ε, ε, μια πολύ σημαντική περιοχή για την Ευρώπη, για μια πολύ σημαντική αποθήκη ύδατος για την Ευρώπη. Είναι πόσιμο νερό Δυστυχώς όμως ε, τώρα την ώρα που μιλάμε μολύνεται. Ε, τα υπόγεια ύδατα κινούνται πολύ πιο αργά από ότι τα επίγεια ύδατα μεταφέρονται όμως ε, με τους ποταμούς. Έχουμε λοιπόν διαρροή των υδάτων αυτών προς τα νότια, προς τα ανατολικά, κάτι που ρηπαίνει πολλά πηγάδια στα γειτονικά χωριά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών που κρίνατε παραδεχτεί την αναφορά μου. Έκτοτε ευτυχώς είχαμε κάποιες θετικές εξελίξεις. Καταρχάς το αρμόδιο Υπουργείο έχει ενημερώσει τους πολίτες σε διάφορες γλώσσες. Ε, είχαμε μάλιστα ε, μία ε, ε, έναν δημόσιο διαγωνισμό, ε, φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί μία τσιμεντένια σαρκοφάγος ε, για να περιοριστεί η κίνηση των υδάτων. Αυτό βέβαια μπορεί να λύσει το πρόβλημα για, τον επόμενο αιώνα. Είναι μια σχετικά προσωρινή λύση. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα που έχουμε κληρονομήσει, την υπόγεια ρήπανση τη ρήπανση των υπόγειων υδάτων που ακόμη δεν έχουν καθαριστεί. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό θέμα και ε, θα πρέπει να γίνει. Γι' αυτό με όλο το σεβασμό σας παρακαλώ να ε, διατηρήσετε ανοιχτή αυτή την αναφορά, διότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει περισσότερη προσοχή στο πρόβλημα αυτό που επισημαίνω στην αναφορά μου. Η επίλυση του προβλήματος αυτού θα απαιτήσει χρόνο. Αρκετές ε, κυβερνήσεις ε, θα δούμε στο μεταξύ. Όλες θα πρέπει να εξετάσουν το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να ασκηθεί πίεση από πλευρά των Βρυξελών για να βοηθηθούν τα χωριά αυτά, ώστε να μπορέσουν να ανακτήσουν το πόσιμό του είδωρ. Πρόκειται για υδάτινα αποθέματα, πολύτιμα για μας. Σας ευχαριστώ πολύ, η κυρία Μαρκεταμπέμοβα από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, αναφέροντα για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Να σας ενημερώσω στο τελευταίο ανακοινωθέν της ε, Επιτροπής ε, του Μαΐου του 2018 θεωρήσαμε ότι οι Σλοβακές Αρχές εργάζονται με κατεύθυνση την επίλυση ε, του προβλήματος των υπογείων υδάτων, ε, κάτι που επιβεβαιώνεται από το δεύτερο σχέδιο για τα ύδατα του Δούναβη. Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας περί υδάτων θα ε, δημοσιευτεί μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, πολύ σύντομα δηλαδή. Παρακολουθούμε την περιοχή Ε, και ο υδροφόρος ορίζοντας ε, θεωρείται ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση, δεν θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχουν ε, κάποια σημεία παρακολούθησης που έχουν δημιουργηθεί, όπου εξετάζεται η περιεκτικότητα σε χημικά των υδάτων. Αυτό είναι μόνο ένα από τα κριτήρια για αξιολόγηση της κατάστασης. Πάντως ε, θεωρείται ότι τα υπόγεια ύδατα βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η αξιολόγηση των ε, σχεδίων ε, για τις λεκάνες των ποταμών φαίνεται να είναι ικανοποιητική. Παρακολουθούμε τα προγράμματα αυτά και ξέρουμε ότι οι προθεσμίες που έδωσαν αρχικά οι σλοβακικές αρχές δεν τηρήθηκαν, παρότι συνεχίζεται η προσπάθεια. Η σχετική διαδικασία ξεκίνησε το 2018 και το Δεκέμβριο του 2018 είχαμε μια αρνητική απόφαση. Αυτό είναι ανησυχητικό. Διάφορες προσφυγές απορρίφθηκαν Υπάρχει όμως η δυνατότητα άσκησης έφεσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει ε, δύο ενστάσεις ε, σχετικά με τη διαδικασία μελέτης αντικτύπου και την οδηγία περί υδάτων. Ε, ισχυρίστηκαν οι υποβάλλοντες ότι η κυβέρνηση της Σλοβακίας δεν ε, συμμορφώνεται με την οδηγία περί υδάτων. Θα επιμείνουμε στη συμμόρφωση με την νομοθεσία, διότι αυτό είναι μία από τις ε, προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να ε, επιθεωρήσει την κατάσταση. Θα εξετάσουμε όμως τα παράπονα σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης με την οδηγία περί υδάτων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος ευρωβουλευτής που θέλει να πάρει το λόγο. <coughs> Θα συνεχίσετε τις έρευνες. Είναι σημαντική οδηγία αυτή και πάρα πολλές χώρες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει εν πάση περιπτώσει την ευθύνη της ως θεματοφύλακα της συνθήκης. Και όχι μόνο η Επιτροπή αλλά και οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων. Νομίζω ότι οι δηλώσεις Κοιτάξτε, η Επιτροπή είναι αυτή η οποία θα πρέπει να ελέγξει ότι ε, οι κυβερνήσεις βρίσκονται στο επίπεδο των απαιτήσεων που υπάρχουν. Να ακούτε καλύτερα τι λέω, λέει η κυρία Ούκεν. Ε, λοιπόν, παραμένει λοιπόν. Θα αποσταλεί στις αρμόδιες αρχές για να υπάρξει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε σχέση με τη συγκεκριμένη οδηγία. Ο κύριος Όρος Σας ευχαριστώ για την απόφασή σας, τίποτα περισσότερο. Sorry. is 443 from 2018. 443 του 18, Μάρκο Τζοβανέλη από την Ιταλία. Ο αναφερόμενος δεν είναι παρόν. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την κυρία Τσαμόρα Εσκριμπάνο, από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας, να μας μεταφέρει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Θα ξεκινήσω την παραμβασή μου με τις νομικές πλευρές της υπόθεσης. Όπως γνωρίζετε στο άρθρο 13 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσει για την ευημερία των ζώων το άρθρο αυτό δεν αφαρμόζεται στις περιοχές όπου δεν υπάρχει νομική βάση για την εναρμόνιση των ε, συνθήκων ζωής, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση όπου έχουμε ε, με ε, επίσης τα οικόσιτα ζώα και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια των κατοικιδίων και αδέσποτων ζώων επίσης. Είναι υπό επεξεργασία προτάσεις νομοθετικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο να προσθέσω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει πλήρως και έχει ξεκινήσει ορισμένες πρωτοβουλίες σχετικές με το αντικείμενο της συγκεκριμένη οδηγίας. Καταρχάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια της Διεθνούς Συνεργασίας για την Ευημερία των Ζώων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στις προσπάθειες για τον έλεγχο των αδέσποτων σκύλων και ε, αναζητείται ο καλύτερος τρόπος έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι συστάσεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει. Υποστηρίζεται επίσης κάθε προσπάθεια για την ευημερία των ζώων της συγκεκριμένης πλατφόρμας, όπως επίσης και προβλέπεται βοήθεια προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης για τη σωστή εφαρμογή των διεθνών κανόνων. Μια άλλη πλευρά ε, συμμετοχής της Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πλατφόρμα για την ευημερία των ζώων που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017. Είναι μια πρωτοβουλία εθελοντικού χαρακτήρα για την υγεία και την ευημερία των ζώων τα οποία γίνονται αντικείμενο εμπορίου και ζητείτε να υπάρξει κατάρτιση καταλόγου όλων αυτών των ζώων στα διάφορα κράτη-μέλη. Προετοιμάζουμε επίσης ε, και ε, ένα δίκτυο ελέγχου για τις πωλήσει online γάτων και σκύλων. Και ήδη τα κράτη-μέλη έχουν αρχίσει να ανταποκρίνονται. Συλλέγουμε λοιπόν πληροφορίες και θα δώσουμε τις πληροφορίες αυτές, αλλά είπαμε ότι στην παρούσα φάση δεν έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε προτάσεις νομικής, ε, ε, ε, νομικής φύσης, δεσμευτικής φύσης, αλλά είμαστε σε μόνιμη επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, οι συνάδελφοι έχουν το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, στην αναφορά αυτή καταγγέλουμε για μια ακόμη φορά την έλλειψη που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με την προστασία και τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων. Είναι σαφές και αυτό το αποδεικνύει το Ευρωβαρόμετρο ότι το 54% των ε, Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει με καλύτερο τρόπο, λέει η κυρία Εύη, τα ζώα συντροφιάς και τα οικόσιτα τα γενικά ζώα. Οι πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν προχωρήσει όσο χρειάζεται και στα πλαίσια της στρατηγικής για την ευμερία των ζώων 12-15 και έχουν καταγγελθεί επίσης ε, και οι ελλείψεις που υπάρχουν από ε, τη μελέτη που κυκλοφόρησε μετά από παραγγελία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δεν θα πρέπει να θεωρούνται αντικείμενα, αλλά θα πρέπει να αναγνωριστούν όπως ακριβώς αναγνωρίζονται και στα πλαίσια της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επαναλάβω ότι ελείπουν στην παρούσα φάση κάποιοι κανόνες ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. ελείψη νομικής φάσης δεν είναι σωστό να πούμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα. Σαν παράδειγμα το θέμα των αδέσποτων είναι ένα θέμα δημόσιας υγείας. Είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, θα έλεγα, η ιστορία με τα δέσποιτα ζώα. Είναι σαφές ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει ακόμα πάρει διαρθρωμένη μορφή και σε καμία περίπτωση δεν είναι ιδιαίτερος δεσμευτική. Και υπάρχει και το πρόβλημα Εμπορία παράνομη σκύλων κυρίω, αλλά όχι μόνο και άλλων ζώων, απαιτούνται ε, μέτρα για την αντιμετώπιση της τρέβλωσης του ανταγωνισμού, γιατί δυστυχώς το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ελείπουν νομοθετικά μέτρα. Πρέπει να συμπληρωθεί, εν πάση περιπτώσει, η ελείπουσα νομοθεσία μέχρι τώρα να διασφαλιστεί η συνέχεια και με άλλες ε, αναφορές τις οποίες έχουμε αποφασίσει να κρατήσουμε ανοιχτές. Ε, τα των αδέσποτων της Βουλγαρίας σαν παράδειγμα μας έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και είναι σαφές ότι ε, στα πλαίσια της επόμενης κοινοβουλευτικής περίοδου και να στείλουμε την αναφορά και στον με μια μικρή πρόσκληση. Τελειώνω εδώ ζητώντας να επικυρώσει ε, και την ε, σύμβαση την διεθνή ε, για την προστασία των ζώων συντροφίας. Γιατί δεν τις έχει επικυρώσει ακόμα παρά μόνο λίγα μέλη το έχουν κάνει αυτό. Και επίσης θα πρέπει να ενημερωθεί και από την ομάδα τη ΜΙΚΤΗ για την ευημερία των ζώων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να διαβιβαστεί στον Επίτροπο Ανδρουκαΐτης. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραβιάζει πάντα το άρθρο 13 της Συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Ε, μιλάμε για την ευημερία των ζώων. Ποια είναι λοιπόν η διαφορά ανάμεσα στον ζώων της κτηνοτροφίας και των ζώων συντροφιάς. Θα πρέπει λοιπόν να μας ενδιαφέρει η ευημερία όλων των ζώων και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το, να το λάβει αυτό υπόψη της. Και όσον αφορά το άρθρο 13 της Συνθήκης της Λισαβόνας, γνωρίζουμε ότι έχει δημιουργηθεί εδώ ένα μεγάλο κενό. Γιατί δεν το κλείνουμε αυτό και γιατί δεν αναδιατυπώνουμε το άρθρο 13. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Ε, δεν ε, είπε κανείς ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί ποτέ η συνθήκη της Λισαβόνας. Και όπως είπε και η ε, συνάδελφος Εύη, τα ε, αδέσποτα ζώα είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στην Ρουμανία το είδα αυτό, υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχουν πολλά τραυματισμένα παιδιά, διότι Πολύ συχνά ε, σπάνε στο ξύλο στο δρόμο τα αδέσποτα ζώα και ε, πολλά παιδιά έχουν πάθει ψυχολογικό, ψυχολογικό τραύμα από αυτό. σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα δεν είναι αδέσποτα ζώα, απλά δεν έχουν βρει τον ε, ιδιοκτήτη τους. Θα πρέπει λοιπόν να διαβάσουμε το θέμα αυτό στον Επίτροπο Άνδριου Καΐτης και στον τομέα αυτό να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμεθα. Δεν έχει νομική βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε όμως κάλλιστα να στείλει συστάσεις στα κράτη-μέλη σχετικά με το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάντλ, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά ότι υπάρχει το πρόβλημα αυτό και ότι μάλιστα είναι δυσανάλογα μεγάλο το πρόβλημα στην Ιταλία. Καταλαβαίνω επίσης ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Φυσικά πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσονται ε, οι ευρωπαϊκές ε, συνθήκες αλλά όχι να δώσουμε στην Ευρώπη αρμοδιότητες που δεν έχει σήμερα και που δεν θα πρέπει να έχει, αλλά ε, ήδη στις 30 Νοεμβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα στο θέμα αυτό, κάτι που έχουμε πει άλλωστε στον αναφέροντα, γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να κλείσει η αναφορά. Ωραία, να στείλουμε λοιπόν επιστολή στον Επίτροπο. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Και δεύτερον, ζητήθηκε να σταλεί επιστολή στην ε, αρμόδια ομάδα για την ευημερία των ζώων. Και έχουμε τώρα έτοιμα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και έχουμε ένα έτοιμα να κλείσει η αναφορά. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν έχει αρμοδιότητες στον τομέα αυτών. Αφού λοιπόν τα κάνουμε όλα αυτά, πιστεύετε ότι πρέπει να κλείσουμε την αναφορά. Ναι. Η κυρία Εύη. Εγώ θα προτιμούσα να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Μια και έχουμε και άλλες αναφορές για το ίδιο θέμα. Και μάλιστα ζητήσαμε στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία να προβλεφθούν και επισκέψεις. Για λόγους λοιπόν συνέπειας και ίσης μεταχείρισης των διαφόρων αναφορών, καλό είναι να κρατήσουμε και αυτή την αναφορά ανοιχτή, όπως και τις προηγούμενες. Είμαι έτοιμη να δεχτώ αυτή την θέση και να κρατήσω ανοιχτή την αναφορά. Συμφωνούμε? Την κρατάμε ανοιχτή. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Τελευταία αναφορά. The last petition for today is... Uh, Τελευταία αναφορά είναι η 0152 του 2017 ο αναφέροντας είναι ο Μάρκο Τζοβανέλη από την Ιταλία. Ο αναφέροντας δεν είναι παρόν, φυσικά, όπως είπαμε και πριν. Μιλάμε για τον Ιταλικό Λίκο. Ο Μάρκο Τσιπριάνη θα θέλαμε να μας πει ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά Υποβλήθηκε το 2017 και αφορούσε το σχέδιο της Ιταλίας για τη διατήρηση και διαχείριση του λύκου της Ιταλίας, του Ιταλικού λύκου. Η αναφορά αφορούσε, ήταν κατά ενός από τα μέτρα του σχεδίου, της δυνατότητα δηλαδή, να εφαρμοστεί η παρέκκληση με βάση την οδηγία για τα οικοσυστήματα, τα ενδιατήματα, για να επιτρέψουμε ε, περιορισμένη θανάτωση μεμονωμένων λύκων σε ορισμένες, υποορισμένες προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή το σχέδιο αυτό δεν έχει υιοθετηθεί, δεν έχει εφαρμοστεί. Η Κομισιόν παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ιταλία και αυτό το σχέδιο συζητήθηκε μεταξύ των διαφόρων φορέων. Η εθνική κυβέρνηση και οι περιφερειακές αρχές το συζήτησαν. Το διαπραγματεύτηκαν, το αναθεώρησαν το ανέβαλαν, το ξανααναθεώρησαν. Από τα τελευταία νέα που έχουμε για τον Ιταλικό λύκο, που τα μάθαμε μέσα από το, τις Ιταλικές εφημερίδες πριν από μερικές εβδομάδες, προκύπτει ότι ο Ιταλός Υπουργός Περιβάλλοντος έχει την πρόθεση να υποβάλει το σχέδιο, ε, το σχέδιο αυτό στις περιφέρειες, ούτω ώστε να εγκριθεί. Το προσχέδιο μάλλον αυτό. Ε, και η Κομισιόν καλωσορίζει αυτή την πρόθεση, γιατί κατά την άποψή μας θα ήταν ένα σημαντικό βήμα αυτό για να εφαρμοστεί αυτό που θέλουμε, που είναι ένα πλήρες σύστημα για να διαχειριστούμε τους λύκους χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία και να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα για να βελτιωθεί η παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο, για να βελτιωθεί η καταπολέμηση της παράνομης σφαγής, της παράνομης θανάτωσης των λύκων, ε, συστήματα προστασίας για τα ζώντα ζώα, να, μιλήσουμε, να μειώσουμε τις ε, συγκρούσεις με κάποιους φορείς και να υπάρξει καλή συνύπαρξη. Θα εξακολουθούμε λοιπόν να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα δούμε εάν το σχέδιο αυτό της Ιταλίας θα υιοθετηθεί. Θα δούμε τι είδου τελικό κείμενο θα προκύψει και πώς θα εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, Κύριε Εύη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ικανοποιημένη από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αντιπροσωπεύει αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ιταλία. Η αναφορά την οποία έστειλε ο συγκεκριμένος πολίτης κατήγγειλε το προηγούμενο πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης για την διαχείριση του λύκου που προέβλεπε επίσης και θανατώσεις ελεγχόμενες του συγκεκριμένου ζώου. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο στο νέο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται. Είμαι ικανοποιημένη διότι ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος η άποψή μου είναι ότι κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και έχει παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα το οποίο ακυρώνει την συγκεκριμένη δυνατότητα. Είμαι ικανοποιημένος γιατί στην Ιταλία λόγω της παράνομης ε, θύρας ε, η οποία είναι πάντα ε, διαδεδομένη, θανατώνονται 800 περίπου λύκοι το χρόνο σε ένα πληθυσμό 5.500 ζώων συνολικά και αυτή η κατάσταση, η κατάσταση πρέπει να αποφευθεί με τα νέα μέτρα. Απαιτείται λοιπόν μια κατάλληλη απάντηση, θα ήθελα να ζητήσω όμως να παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη οδηγία γιατί το πρόγραμμα δεν έχει γίνει απόλυτα δεκτό, ε, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να εγκριθεί από τις περιφέρειες, ιδιαίτερα από τις περιφέρειες Μίλια, Ρωμάνια, Τρέντο, Μπολτσάνο, Πεδεμόντιο Γενικά είναι σημαντικό λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη οδηγία έτσι ώστε να υπάρξει απαιτούμενη συνένεση και ζητώ να αποσταλεί η συγκεκριμένη αυτή η αναφορά στις περιφέρειες έτσι ώστε να υπάρξει σωστή ενημέρωση και πίεση γιατί όχι μόνο οι πολίτες, Ιταλοί και Ευρωπαίοι αλλά και η Επιτροπή μας ε, θέλει να αποφύγουμε μια διαχείριση του ζώου που προβλέπει τις επιλεκτικές θανατώσεις. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι το νέο πρόγραμμα για τους λύκους είναι πολύ σημαντικό. Οι πόροι οι οποίοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα χρησιμοποιηθούν μέσω του προγράμματος LIFE θα χρησιμοποιηθούν με πιο σωστό τρόπο και έτσι ελπίζω να καταστούν πρότυπο για άλλα κράτη-μέλη και να μπορέσουμε να πούμε ότι η συμβίωση ανθρώπων και λύκων γίνεται εφικτή μέσω των προληπτικών μέτρων. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που θίγεται το θέμα. Είναι πολύ συγκλονιστικά τα νούμερα που δίνεται, 800 από 2.000. Ο Λύκος έχει πολύ ε, κακή φήμη, όλοι το γνωρίζουν, τρώνε τις γιαγιάδες. Ε, έτσι πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να ξεφορτωθούμε αυτό το τρομερό ζώο. Αλλά να το πω διαφορετικά. Όταν ακούω το τι γίνεται για να προστατεύσει κανείς ε, τα εκτρεφόμενα ζώα, Στη Δανία δεν έχουμε τόσους λύκους, έχουμε όμως την ίδια συζήτηση. Αν έχει κανείς έναν καλό ασφαλή φράχτη, μπορεί να προστατεύσει τα ζώα εκτροφής. Εάν επιμένει κανείς να ξαμολάει τα πρόβατά του, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε όλη τη φύση, δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στα πρόβατα. Στο παρελθόν είχε κανείς βοσκούς και σκυλιά που φιλούσαν τα ζώα. Εάν θέλετε να αμολάτε στη φύση τα ζώα, δεν μπορείτε να ε, περιμένετε από τη φύση να μην είναι φύση και από τα αγρία ζώα να μην είναι αγρία ζώα. Θα ήθελα πολύ να δω το σχέδιο και θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν συμπεριλαμβάνεται ευθύνη των ιδιοκτητών ή περιμένουμε από τη φύση να συμπεριφερθεί ευγενικά. Δεν θα έλεγα ανθρώπινα, διότι εμεί σκοτώνουμε τα ζώα. Αλλά, εν πάση πτώση, περιμένουμε από τα ζώα να μην φερθούν σαν ζώα. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριο Μάντλ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ακούω με ενδιαφέρον τη συζήτηση. Βρίσκω ότι είναι σημαντικό το θέμα, διότι σε πολλά μέρη της Ευρώπης ε, αυξάνεται η πρόκληση των λύκων, διότι αποτελούν κινδυνό για ανθρώπους και ζώα. Είναι σημαντικό να γίνει συζήτηση. Αναφέρθηκαν οι φράχτες που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία, για παράδειγμα ε, για τα εγωπρόβατα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνουν οι επενδύσεις αυτές και τι θα σημαίνουν για ε, την Ήπεθρο δεν πρέπει να προστατεύσουμε μόνο τους λύκους, πρέπει να προστατεύσουμε και τα πρόβατα καθώς ε, και, και άλλα ζώα συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Στην ε, Ιταλία, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει νομοθετική διαδικασία σε περιφερειακό επίπεδο, αυτό είναι σημαντικό, αλλά ε, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει στόχο να στηρίξει ή να σχολιάσει η νομοθετική διαδικασία ε, στα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν στις 31 ε, Οκτωβρίου του 2017 διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει κάποια ε, παραβίαση των κανόνων από την Ιταλική κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν έχει καμία θέση εδώ και πιστεύω ότι θα πρέπει να κλείσει. So we have a problem again. Uh, Υπάρχουν δύο διαφορετικές θέσεις. Αρνείστε, Πρόεδρε, ότι το 2000, το, το Natura 2000 είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα. Υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις. Καλά νέα για αυτό το θέμα. Δεύτερον, ας περιμένουμε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα των Ιταλικών αρχών. For Τι να κάνουμε, ποια είναι η άποψη Εγώ δεν είμαι υπέρ του να κλείσουμε κατά ανάγκη αυτή την αναφορά, αλλά... Κυρία Εύη, ποια άποψη έχετε. Κύριε Πρόεδρε, να πάρω το λόγο. Ακόμα και η Κομισιόν είπε ότι θα εξετάσει τη διαδικασία. Uh, Γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει μέχρι να τελειώσουν όλα. Είμαστε η Επιτροπή Αναφορών. Οι πολίτες μας έχουν εμπιστοσύνη. Θέλουν και χάρη σε εμάς να εφαρμοστεί σωστά η ενωσιακή νομοθεσία. Θα προτιμούσαν να κρατήσουμε ανοιχτή και αυτή την αναφορά, όπως και την προηγούμενη, να έχουμε έτσι το βλέμμα μας εκεί, το νου μας. Ας περιμένουμε να κλείσει η, κοινοβουλευτική διαδικασία, η νομοθετική συγγνώμη, διαδικασία στην Ιταλία και όταν τελειώσει θα κλείσει και η αναφορά αυτή. Γεια Ροσλάβ. Φυσικά θέλουμε να κρατήσουμε τελικά τις αναφορές ανοιχτές, αλλά κάποια στιγμή δουλειά μας είναι να κρατήσουμε ε, αναφορές ανοιχτές όταν είναι αρμοδιότητά μα. Ε, και να έχουμε και μια λογική. Δεν είναι λογικό, α πούμε, κατά όλες τις αναφορές αναφορέ ανοιχτές. Ε, ίσως δεν είναι και τόσο κακή ιδέα να κλείσουμε κάποιε αναφορέ. Εγώ θα προτιμούσα να την κλείσουμε. Νομίζω είναι καλή ιδέα. Όλα... Έχουμε δύο-τρία άτομα από Εάν έχουμε δύο-τρία άτομα από το ΕΛΚ που πάντα θέλουν να κλείνουν τι αναφορέ, θα τι κλείσουμε όλε. Αλλά ήταν σαφέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν εξελίξει στο θέμα αυτό. Είναι θέμα που ενδιαφέρει πολλέ χώρε και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε σωστή απάντηση. Έχουμε κάτι που μοιάζει με πλειοψηφία, αλλά να θυμάστε ότι δεν έχουμε απαρτία. Αλλά αν είναι να το κάνουμε αυτό, να κλείσουμε όλε τι αναφορέ. Δεν υπάρχει πραγματικό λόγο να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Υπάρχει πραγματικό λόγο να την αφήσουμε ανοιχτή. Αν είναι έτσι με δύο ψήφους να κλείνουμε όλες τις αναφορές... Ε, όχι, όχι. Επί της αρχής ε, συμφωνώ με τους συναδέλφους, ε, διότι Πιστεύω ότι είναι σωστή η θέση αυτή. Πρόκειται για μια επιτυχία αναφορά. Έχουμε πολύ σαφείς εξελίξεις, πολύ σαφή βήματα πρόοδου. Αλλά δεν θα ήθελα σύγκρουση τώρα στο τέλος ε, ε, αυτής της ε, συνεδρίασής μας. Ωραία, να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να στείλουμε επιστολή στις Ιταλικές Αρχές, να τους ζητήσουμε νέες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Αυτά για σήμερα. Ωραία μέρα περάσαμε. Εντάξει, ήτανε... είχαμε πολλή δουλειά. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 9. Καλό σας βράδυ.